έχουν πέσει οι τιμές του πετρελαίου και μειώθηκαν επίσης και οι δραστηριότητες, οι οικονομικές δραστηριότητες και οι συνθήκες λειτουργίας της αγοράς. Κατά το 2009 για μερικούς μήνες ήταν αρνητικός ο πληθωρισμός κυρίως λόγω της δυναμικής των τιμών του πετρελαίου και των επιπτώσεων της. Αν αποκλείσουμε την ενέργεια και τις τιμές των τροφίμων, ο πληθωρισμός από τα μέσα του 2008 έχει αρχίσει να πέφτει ιδιαίτερα γιατί μειώθηκε το κόστος της εργασίας αλλά και τα περιθώρια κέρδους. Τον Μάρτιο του 2010 η Ευρωζώνη γνώρισε 1,4 πληθωρισμό και αυτό οφειλόταν κυρίως στις εξελίξεις που αφορούσαν τα τρόφιμα και την ενέργεια. Λόγω της αργής αναθέρμανσης και υψηλότερης απασχόλησης παραμένει βραδία η ανάπτυξη και φέτος. Δεν αναμένονται μεγάλες εξελίξεις για τον πληθωρισμό γιατί θεωρούμε ότι ο στόχος μας μη ε, συγκράτησης τον του πληθωρισμού έχει πετύχει. Αναμένουμε οι επιπτώσεις του πληθωρισμού στις τιμές να δείξουν πόσο αξιόπιστη είναι η πολιτική της ΕΚΤ της τη συγκράτηση των τιμών. Η αξιολόγηση μας δείχνει ότι μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα ισχύουν όλα αυτά διότι Οι δανειοδοτήσεις προς τον ε, ιδιωτικό τομέα μειώθηκαν και προς τα τέλη του περασμένου έτους υπήρξε αρνητική ανάπτυξή τους. Τελικά, οι τελευταίες εξελίξεις στα χρηματοπιστωτικά δείχνουν ότι είναι χαμηλός ο κίνδυνος αύξησης του πληθωρισμού βράχη και μεσοπρόθεσμα. Το Φεβρουάριο του 2010 είχαμε μείον 0,4% πληθωρισμό και παραμένει χαμηλή η ανάπτυξη, γι' αυτό θα παραμείνει χαμηλός και ο πληθωρισμός. Η αρνητική επίσης ανάπτυξη των δανειοδοτήσεων δείχνει ότι τους τελευταίους μήνες οι δανειοδοτήσεις έχουν ωφελήσει κυρίως τους ιδιώτες. Οι διαφορετικές αυτές ε, τιμές ανάλογα με τους τομείς είναι λογικές. Πέρυσι, επειδή δεν υπήρχε υψηλός πληθωρισμός, το Διοικητικό Συμβούλιο μείωσε μεταξύ Ιανουαρίου και Μαΐου κατά 150 βασικές μονάδες σε 1% δηλαδή τις δραστηριότητες του και, τις, ε, και κατέληξαν στα 325 βασικά σημεία. Θεωρεί λοιπόν το Διοικητικό Συμβούλιο ότι τα επιτόκια αυτή τη στιγμή είναι σωστά και η σταθερότητα των τιμών θα διατηρηθεί μεσοπρόθεσμα. Εκτός από τη μείωση των επιτοκίων, το Διοικητικό Συμβούλιο πήρε και άλλα μέτρα στήριξης της δανειοδότησης για να βελτιωθεί η κατάσταση και για να μπορέσουν να συνεχίσουν οι δραστηριότητες αυτές. Τα μέτρα αυτά έχουν πετύχει το στόχο τους. Ιδιαίτερα έχουν μειώσει τα επιτόκια των τραπεζών και έτσι στήριξαν τη χρηματοδότηση και των ιδιωτών και των εταιριών. Γενικά, η επίκαιρη και αποτελεσματική δράση μας σε απάντηση στην κρίση, καθώς και η σταθερή προσήλωση της ΕΚΤ στη διατήρηση της σταθερότητας των τιμών, θεωρούμε ότι μεσοπρόθεσμα έχει πετύχει και στηρίξει την αναθέρμανση της Ευρωζώνης, στην Ευρωζώνη. Θα ήθελα να τονίσω ότι όταν η ΕΚΤΕΝ έκρινε αυτές τις ε, αυτά τα καινοτόμα μέτρα, ήδη είχε στο μυαλό της τη στρατηγική της προοδευτικής μείωσης facing out. Το ευρωσύστημα είχε προβλέψει την προοδευτική μείωση αυτών των έκτακτων μέτρων εφόσον δεν θα χρειαζόνταν πια. Είχε προβλεφθεί ένα χρονοδιάγραμμα που να αποφεύγει οι στρεβλώσεις της αγοράς που θα υπήρχαν αν διατηρούνταν τα έξακτα αυτά μέτρα περισσότερο χρόνο από όσο χρειαζόταν. Το Σεπτέμβριο του 2009 και το Μάρτιο του 10 αποφασίσαμε προοδευτικά να μειώσουμε ορισμένα από τα έκτακτα μέτρα για τη ρευστότητα, τον αριθμό, τη συχνότητα και την οριμότητα μακροπρόθεσμων χρηματοδοτήσεων. Το Μάρτιο αποφασίσαμε να επιστρέψουμε στις κανονικές τριμηνιές χρηματοδοτικές μας λειτουργίες με αρχή αύριο και συνεχίζουμε να χορηγούμε ρευστό στους παράγοντες της αγοράς Και θεωρούμε ότι έτσι διευκολύνουμε τη χορήγηση δανείων στην ευρωπαϊκή οικονομία και στηρίζουμε περαιτέρω ακόμη την αναθέρμανσή της. Βεβαίως, εάν υπάρξουν διαταραχές των τιμών αύξηση τους, δηλαδή το Διοικητικό Συμβούλιο θα πάρει τα μέτρα που χρειάζονται. Τώρα, κυρία Πρόεδρε, θα γυρίσω στα φαραλαγικά. Ο προϋπολογισμός της Ένωσης επλήγει ιδιαίτερα πέρυσι από την κρίση και το φορολογικό κίνητρο καθώς και τα κυβερνητικά μέτρα χρειάζεται έγιναν απαραίτητα. Το Ευρωστάτ υπολόγισε ότι κατά μέσο όρο το, έλλειμμα, το κυβερνητικό έλλειμμα αυξήθηκε από 2% του ΑΕΠ το 8 σε 6,3% το 9. Από τις 16 χώρες της Ευρωζώνης, 13 ήδη έχουν υπερβολικό έλλειμμα. Και φέτος όλες οι χώρες της Ευρωζώνης θα έχουν έλλειμματα πάνω από το προβλεπόμενο 3% του ΑΕΠ. Τα προγράμματα σταθερότητας δεν προβλέπουν βελτίωση πριν από το 2011 με 12 και το μέγεθος της, ε, του προβλήματος στα δημοσιονομικά που βασίζεται στα ενημερωμένα προγράμματα σταθεροποίησης δείχνει ότι ο μέσος όρος του ελλείμματος θα αυξηθεί κατά 21% σε σύγκριση με πέντε χρόνια πριν. Οι δημοσιονομικές ανισότητες, ανισορροπίες λοιπόν θα συνεχίσουν θα διατηρηθούν. Τα προβλήματα αυτά ήταν ιδιαίτερα οξέα σε ορισμένες χώρες, την Ιρλανδία, την Ελλάδα και την Ισπανία, που είχαν διψήφιο έλλειμμα. Οι αλλαγές στον προϋπολογισμό της Ελλάδας, ή μάλλον τα δεδομένα που αφορούσαν τον προϋπολογισμό της Ελλάδας, έδειξαν σοβαρό έλλειμμα και προκάλεσαν σοβαρές αντιδράσεις της αγοράς. Μετά από τα μέτρα που έλαβαν οι ελληνικές αρχές το Μάρτιο του 2010, τα οποία δέχεται η ΕΚΤ, θεωρούμε ότι πρόκειται για πιστική πολιτική για βελτίωση των δημοσιονομικών της χώρας αυτής. Όλα αυτά τα μέτρα πρέπει να εφαρμοστούν βέβαια εγκαίρως. Παρά όμως την προσήλωση της ελληνικής κυβέρνησης στα μέτρα αυτά και τις δηλώσεις των αρχηγών κρατών κυβερνήσεων της Ευρωζώνης της 25ης Μαρτίου και του Eurogroup συνέχισαν οι πιέσεις και εντατικοποιήθηκαν πρόσφατα. Είναι βασικό το οικονομικό πρόγραμμα που προετοιμάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η ΕΚΤ, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και οι ελληνικές αρχές να προβλέψουν και δομικές αλλαγές που να λύνουν τις, τους λόγους της δημιουργίας του προβλήματος της Ελλάδας έτσι ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη σταθερότητα των δημοσίων οικονομικών και να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα της χώρας. Γενικότερα τώρα υπάρχουν ανησυχίες ότι η διατήρηση των δημοσιονομικών τέτοιων ανάλογων προβλημάτων θα υπονομεύσει γενικότερα στην Ευρώπη την οικονομική ανάπτυξη και τη δημοσιονομική χρηματοδοτική σταθερότητα. Όπως έχουν τώρα τα πράγματα, το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης που δημιουργήθηκε για να διατηρηθεί η ανάπτυξη αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη του πρόκληση από, τη, από το 1997 που δημιουργήθηκε. Γι' αυτό είναι απαραίτητο τώρα όλες οι χώρες της Ευρωζώνης να εφαρμόσουν αυστηρά το σύμφωνο. Τώρα από θετικά, θετικό είναι ότι όλες οι χώρες της Ευρωζώνης που έχουν υπερβολικό έλλειμμα έχουν προβλέψει να το διορθώσουν μέσα στα χρονοδιαγράμματα του Συμβουλίου. Και επίσης ενθαρρυντικό είναι ότι τα περισσότερα από αυτά τα προγράμματα προβλέπουν μείωση των κυβερνητικών δαπανών, γιατί τα στοιχεία δείχνουν ότι αυτό είναι ο αποτελεσματικότερος τρόπος για μείωση των ανισοτήτων αυτών, των ελλημάτων. Σε πολλά όμως από αυτά τα σταθεροποιητικά προγράμματα δεν τονίζεται αρκετά σε ορισμένες περιπτώσεις η πραγματική κατάσταση αλλά μπορούμε να πούμε ότι τα προγράμματα αυτά είναι υπερβολικά αισιόδοξα. Εμείς δεχόμαστε τη δήλωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 25ης Μαρτίου του Ευαγγελισμού δηλαδή ε, για ενδυνάμωση του υπάρχοντος θεσμικού συστήματος για καλύτερη δημοσιονομική πειθαρχία η δημιουργία μιας ειδική ομάδας task force για να βρεθούν, να εξεταστούν όλες οι δυνατές λύσεις για το πρόβλημα αυτό είναι κάτι το θετικό, ιδιαίτερα δε είναι βασικό να βελτιωθούν, να δοθούν περισσότερα κίνητρα για τις εθνικές αρχές ώστε να εφαρμόσουν προγράμματα εγκαίρως που να σταθεροποιούν τα δημοσιονομικά τους και να διασφαλίσουν ότι η οικονομική επιτήρηση ή εποπτεία θα καταλήξει σε αποτελεσματική πολιτική που να λύνει τα διαρθρωτικά προβλήματα και να αυξάνει την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών οικονομιών. Κυρία Πρόεδρε, τώρα νομίζω ότι θα καταλήξω με θέματα που αφορούν την επιτήρηση και την εποπτεία. Σε ό,τι αφορά την μεταρρύθμιση στα ρυθμιστικά θέματα όπως καθορίστηκε από τους ηγέτες των G20 <clears throat> έχουν γίνει ευρείες και σημαντικές εργασίες ή συνεχίζονται ακόμα αυτές οι εργασίες. Δεν πρέπει όμως να χαλαρώσουμε την προσοχή μας. Είναι απαραίτητο η ορμή η οποία έχει δημιουργηθεί για μεταρρύθμιση να μην μειωθεί. Είναι πολλά ακόμα αυτά τα οποία πρέπει να πράξουμε. Καταρχήν είναι απαραίτητο τα σχέδια μεταρρύθμισης να οδηγήσουν σε μια εναρμονισμένη παγκόσμια μορφή ρύθμιση, ένα πλαίσιο ρύθμιση σε παγκοσμίο επίπεδο. Δεύτερον, είναι κατεπίγουσα προτεραιότητα οι προτάσει τη Επιτροπή Βασιλεία για τι κεφαλουχικέ ε, απαιτήσει, τα πρότυπα ρευστότητα και τα αντισταθμιστικά μαξιλάρια μέσα σε εισαγωγικά να μπορέσουν να εφαρμοστούν μέχρι το τέλο του 2010. Πρέπει να εξασφαλίσουμε επίση ότι το ρυθμιστικό αυτό πλαίσιο αντιμετωπίζει όλα τα συστημικά σημαντικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και αντιμετωπίζει και τα προβλήματα ηθικού κινδύνου που συνάπτονται με αυτά τα ιδρύματα. <clears throat> Μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι βελτιώσεις της οδηγίας για την κεφαλογική επάρκεια θα πρέπει να εγκριθούν ταχαίως και μία έγκριση της οδηγίας για εναλλακτικά ταμεία επενδύσεων επίσης πρέπει να εγκριθεί. Σε ό,τι αφορά την δημιουργία του νέου εποπτικού πλαισίου μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα είναι απαραίτητο η νομοθετική διαδικασία για τις προτάσεις της Κομισιόν να μπορέσει να συμπληρωθεί το ταχύτερο δυνατό. Και επίση ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι να μπορέσουν να καταλήξουν μια συμφωνία σε σχέση με ένα νομικά δεσμευτικό κείμενο, ώστε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου και οι Ευρωπαϊκέ Εποπτικέ Αρχέ να λειτουργούν ήδη από την 1η Ιανουαρίου του 2011 δεν θα πρέπει να διακινδυνεύσουμε να χάσουμε την ορμή μας στην πορεία αυτή μεταρρυθμίσεων. Θέλω να τονίσω επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει προχωρήσει σημαντικά για να μπορέσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου να λειτουργήσει σωστά από τη στιγμή που θα θεσπιστεί. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η υποστήριξη η οποία θα πρέπει να δοθεί από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στο Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου και η αμοιβαίοι δεσμοί δεν θα επηρεάσουν την ανεξάρτητη λειτουργία αυτού του Συμβουλίου και την επίτευξη των στόχων του που καθορίζονται σαφώς πάνω της ευρωπαϊκή Τράπεζας που καθορίζονται σαφώς στις συνθήκε. Ο στόχος μας παραμένει η διατήρηση της σταθερότητας τιμών και η διαχείριση της κοινή νομισματικής πολιτικής έχει αυτό σαν απότερο στόχο. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και οι Εθνικέ Κεντρικέ Τράπεζε διατηρούν ακόμα την ανεξαρτησία του σε ό,τι αφορά του στόχου που του αποδίδει η συνθήκη. Επομένω δεν μπορεί να υπάρξει και δεν θα υπάρξει <clears throat> καμία δυνητική σύγκρουση μεταξύ τη διαχείριση τη νομισματική πολιτική από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με στόχο τη διατήρηση τη σταθερότητα τιμών και την εκτέλεση καθήκοντων που έχουν να κάνουν με την διατήρηση και την επίτευξη χρηματοπιστωτική σταθερότητα οι συστάσεις της Κεντρικής Τράπεζας δεν αφορούν τον τρόπο με τον οποίο θα εφαρμοστεί η λειτουργία κεντρικών τραπεζών εκτός της ζώνης του ευρώ. Συγχρόνως, η μακροπολιτική εποπτεία μπορεί να διευκολύνει την διαχείριση και την ε, λειτουργία της νομισματικής πολιτικής με το να προβλέψει συστημικούς κινδύνους και να μετριάσει τα αποτελέσματά τους εάν παρουσιαστούν τέτοιες κρίσεις. Πρώτο κλείσω λοιπόν, θέλω να τονίσω και πάλι ότι μια έγκαιρη και συνεκτική εφαρμογή του εποπτικού και ρυθμιστικού πλαισίου αυτού και των μεταρρυθμίσεών του, ιδίω η δημιουργία ενό νέου πλαισίου για μακροπροληπτική εποπτεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα συμβάλλει τα μάλα στο να περιορίσουμε του συστημικού κινδύνου και στο να ενισχύσουμε την ανθεκτικότητα του ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού συστήματο. Για την ΕΚΤ είναι μεγάλο προνόμιο το γεγονό ότι μα έχετε επιφορτήσει με αυτό το τόσο σημαντικό ρόλο σε ό,τι αφορά τη μακροπροληπτική εποπτεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρά το γεγονός ότι έχουμε ενώπιόν μας πολλές προκλήσεις και ένα δύσκολο καθήκον, εγώ έχω κάθε εμπιστοσύνη ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε συνεργασία με τις Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες και όλα τα άλλα μέλη της, του Συμβουλίου Τραπεζών στην Ευρώπη θα μπορέσει να φέρει σε πέρα σε αυτό το στόχο. Κύριε Πρόεδρε, έντιμα μέλη της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αυτή ήταν η παρουσίασή μου <clears throat> ενώπιόν σα και είναι η τελευταία φορά που έρχομαι ενώπιόν σα ω αντιπρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Θέλω να λεφτά αυτή την ευκαιρία να σε ευχαριστήσω για την τόσο εμπλουτιστική και επικοδομητική ανταλλαγή απόψεων που είχα μαζί σα όλα αυτά τα χρόνια. Έχω εκτιμήσει ιδιαίτερα τη συνεργασία μαζί σα και τον καρποφόρο διάλογο με την Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σα ευχαριστώ λοιπόν πάλι για την προσοχή σα και φυσικά είμαι στη διάθεσή σα για τα ερωτήματά σα. Uh, Ευχαριστώ, κύριε Παπαδήμου. Τα χειροκροτήματα δείχνουν ότι τα αισθήματα είναι αμοιβαία. Δεχόμαστε ότι πράγματι ήταν πολύ καλή η σχέση σας με αυτή την Επιτροπή. καθώς και με τον Πρόεδρο και τους άλλους αντιπροέδρους. Πάμε στις ερωταπαντήσεις. Να σας πω ποιος είναι στον κατάλογο, ούτω ώστε εκείνοι που θέλουν να μιλήσουν σηκώ το χέρι τους γρήγορα, να μην ανακαλύψω ότι έχω το τελευταίο δεκάλεπτο 20 άτομα. Αυτά είναι τα πρώτα ονόματα. Άλλος που θέλει το λόγο. Okay, well, go first to Wolf Klintz. Ο Wolf Klintz είναι ο πρώτος. Κύριε Αντιπρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το τελευταίο σημείο που αναφέρατε είναι και το πρώτο το οποίο εγώ θα ήθελα να θίξω, λέει ο κ. Κλίντς. Μια στιγμή ο ομιλητής μιλάει πολύ μακριά από το μικρόφωνο, μπορεί να το φέρει πιο κοντά στο... Λειτουργεί το σύστημα. Ναι. Κύριε Αντιπρόεδρε, το τελευταίο σημείο που θίξατε είναι το πρώτο το οποίο εγώ θα ήθελα να αναφέρω και εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω για την εργασία σας, για την ε, συμβολή σας στην ε, επίτευξη σταθερότητα στον χώρο του ευρώ. Εσείς παίξατε ένα προεξάρχοντα ρόλο για την εισαγωγή του ευρώ και τη σταθερότητα και ήσασταν πάντα έτοιμος να συναντηθείτε και εδώ και στη Φραγκφούρτη με τους εκπροσώπους του Κοινοβουλίου. Γι' αυτό σας ευχαριστώ. Έχω τρία σημεία στα οποία θέλω να αναφερθώ τώρα. Πρώτα απ' όλα για την κρίση στην Ελλάδα. Δεν αποκλείεται αυτή τη στιγμή ότι το πακέτο διάσωσης θα, θα πρέπει να συνδυαστεί με μία μείωση των απαιτήσεων των πιστωτών αυτή τη στιγμή. Είναι πολλοί από αυτού του πιστωτέ, βέβαια Ευρωπαϊκέ Τράπεζε και Γαλλικέ και γερμανικέ τράπεζε, οι οποίε έχουν διψήφια δισεκατομμύρια δάνεια προ την Ελλάδα. Αν αυτέ, λοιπόν οι τράπεζε δεχτούν κάποια μείωση των απαιτήσεών του παραδείγματος χάρη σε επίπεδο 30 ή 40%, αυτό θα οδηγήσει τι τράπεζε αυτέ πάλι σε δυσκολία. Βλέπετε να υπάρχει πραγματικά ένα κίνδυνο ότι μέσα από όλα αυτά θα προκύψει μια δεύτερη κρίση στον τραπεζικό τομέα. Αυτό είναι το πρώτο μου ερώτημα. Δεύτερο ερώτημα. Στη χώρα μου, στη Γερμανία, υπάρχουν κάποιοι οικονομολόγοι οι οποίοι λένε ότι αυτό το οποίο αναμένεται από την ε, Ελλάδα, το πακέτο αναδιάρθρωσης, περιλαμβάνει τον κίνδυνο ότι θα προκύψει από μια οικονομική κρίση μια βαθιά ύφεση. Αυτό δεν είναι δική μου άποψη. Αλλά αν θυμηθείτε την ε, πολιτική του κυρίου Μπρίνινγκ, του τελευταίου καγκελαρίου στην Δημοκρατία της Βαϊμάρης μετά τον Εθνικό Σοσιαλισμό, αυτό το οποίο είχε κάνει ο Μπρίνινγκ ήταν ότι ε, έκανε ριζικές περικοπές στο δημόσιο τομέα και με τον τρόπο αυτό οδήγησε στην βαθιά ύφεση που <clears throat> έπληξε τότε τη Γερμανία. Επίσης, το θέμα του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, που είναι δεσμευτικό. Μήπως πρέπει να βρει ένας τρόπο να υπάρξει λύση για το γεγονό ότι έχουμε μια κοινή πολιτική στο νομισματικό τομέα, αλλά δεν έχουμε μια κοινή δημοσιονομική πολιτική. Μήπω θεωρείτε ότι αυτή, αυτό το σύμφωνο σταθερότητα είναι ανεπαρκέ. Και αυτό όχι μονάχα επειδή υπάρχουν πια πολύ συχνά παραβιάσεις του Συμφώνου Σταθερότητος, αλλά γιατί ένα σημαντικό στοιχείο το οποίο είναι απαραίτητο για τη σταθερότητα, δηλαδή το στοιχείο της ανταγωνιστικότητας, ελείπει από το Σύμφωνο σταθερότητας. Βλέπουμε χώρες όπως η Ισπανία, η οποία δεν είχε πρόβλημα στον προϋπολογισμό τη λίγο πριν από την κρίση, <clears throat> αλλά λόγω της κατάρρευση του κατασκευαστικού τομέα και του, των συναφών οικονομικών κλάδων βρέθηκε σε μια πραγματική κατάσταση μεγάλων ελλημάτων λόγω της απώλειας της ανταγωνιστικότητας. Θα ήθελα με μεγάλη, μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσω πώς θα προτείνατε εσείς να επιληθεί το πρόβλημα αυτό. Uh, Νομίζω ότι θα πρέπει να ακολουθήσω, να μαζέψω κάποιες ερωτήσεις και μετά να απαντήσετε. Η Άννη έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Αντιπρόεδρε για την πολύ περιεκτική και ενδιαφέρουσα εισήγησή σας. Έχω δύο σύντομα ερωτήματα να σας θέσω. Το πρώτο αφορά στις διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη αυτή τη βδομάδα ε, ανάμεσα στην ε, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την Ευρωζώνη, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και τις ε, ελληνικές αρχές ε, για την ε, οριστικοποίηση της συμφωνίας που δώσει τη δυνατότητα στην ενεργοποίηση του μηχανισμού υποστήριξης. Ήθελα να σας ρωτήσω ποιος είναι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σε αυτές τις διαπραγματεύσεις αφενός και αφετέρου ποιο συγκεκριμένο ρόλο βλέπετε στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μέσα στα πλαίσια του μηχανισμού υποστήριξης. Το δεύτερο ερώτημα είναι γενικότερο, αφορά στα όσα μας είπατε για τα δημοσιονομικά προβλήματα στην Ευρωζώνη γενικότερα, στο πολύ εντυπωσιακό ε, συμπέρασμα ότι 13 από τις 16 χώρες μέλη της Ευρωζώνης έχουν σήμερα ε, προβλήματα ε, δημοσιονομικής φύσεως. Αναφερθήκατε ασφαλώς ιδιαίτερα στην ελληνική περίπτωση, στα μέτρα που έχουν εξαγγελθεί και ήδη εφαρμόζονται από τις ελληνικές αρχές. Τα χαρακτηρίσατε μάλιστα φιλόδοξα αλλά αναγκαία και υπογραμμίσατε ότι ε, παρά τα μέτρα αυτά η πίεση από την πλευρά των αγορών συνεχίστηκε και μάλιστα τις τελευταίες εβδομάδες ε, διευρύνθηκε. Ήθελα να σας ρωτήσω λοιπόν ε, πού αποδίδετε εσείς αυτή την συνεχιζόμενη και εντυνόμενη πίεση από την πλευρά των αγορών. Αν θεωρείτε δηλαδή ότι εξηγείται από την καχυποψία, την έλλειψη εμπιστοσύνη από την πλευρά των αγορών απέναντι στα μέτρα που έχουν εξαγγελθεί ε, και ήδη έχουν αρχίσει να εφαρμόζονται στην Ελλάδα ε, και εάν θεωρείτε ότι αυτή η πίση αποσκοπεί ε, έχει ως στόχο δηλαδή μόνο την Ελλάδα ή γενικότερα τη ζώνη του ευρώ και κλείνω αμέσως υπάρχει περίπτωση κύριε Αντιπρόεδρε να αναθεωρήσετε, να επανεξετάσετε την πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που αφορά ε, στο γεγονός ότι δεν ε, είναι αποδεκτό να δανείζει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα απευθείας κράτη-μέλη αλλά μόνο εμπορικές τράπεζες με αποτέλεσμα να εντείνεται ε, η κερδοσκοπία σε βάρος εθνικών ομολόγων. Ευχαριστώ πολύ. Περιμένουμε να τελειώσει η διερμηνία. Φίλιπ. Ευχαριστώ κύριε Παπαδήμου. Ευχαριστώ για την ε, παρουσίαση και για την παρουσία σας εδώ. Σαν πράσινη, σεβόμεθα, εδώ είμαι, σεβόμεθα λέω την, Ευρωπαϊκή, την εξαρτησία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Θέλουμε να δούμε το ίδιο επίπεδο ανεξαρτησίας και των πολιτικών όταν αποφασίζουν τη δράση που θα αναλυθεί. Το λέω συχνά στην Επιτροπή αυτή ότι όποτε τονίζει η ΕΚΤ την ανάγκη για φορολογική ενοποίηση, δηλαδή αντιμετώπιση των οικονομικών μέσω αντιμετώπιση των δαπανών, είναι μια πολιτική δήλωση αυτή. Αυτό που είπατε σας βγάζει εκτός της εντολής σας. Είναι πολιτική απόφαση. Να αποφασίσουμε δηλαδή πώς θα πετύχουμε τον κοινό στόχο της οικονομικής υγείας. Συμφωνούμε μαζί σας. Δεν θέλουμε να έχουμε τεράστια ελλείμματα, είναι ανθυγινό και μη βιώσιμο. Αλλά πώ θα το πετύχουμε αυτό, αυξάνοντα τα έσοδα ή μειώνοντα τι δαπάνε, αυτό δεν είναι δική σα δουλειά. Αυτή είναι δική μα δουλειά. Και είμαστε υπόλογοι στου ψηφοφόρου γι' αυτό. Το μέγεθο του δημόσιου τομέα στην οικονομία που δεν είναι δείκτη τη αποδοτικότητα οικονομία. Κοιτάξτε τι γίνεται με την, το, το τομέα τη υγεία. Στη ΣΥΠΑ η υγεία κυρίω είναι του ιδιωτικού τομέα. 16% του ΑΕΠ δαπανάται σε αυτό για ένα αποτέλεσμα που είναι χειρότερο από την Ευρώπη που κατά μέσο όρο το 12% του ΑΕΠ πηγαίνει στην ε, περίθαλψη. Σας παρακαλώ, θα παρότρινα την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αν θέλετε να παραμείνετε ανεξάρτητοι, παρακαλώ να σεβαστείτε την ανεξαρτησία εκείνων που διαμορφώνουν την πολιτική. Αυτοί να αποφασίσουν πώς θα πετύχουν τους στόχους που είναι κοινοί για όλους. Σας ευχαριστώ. Καλώς. Νομίζω ότι συλλέξαμε κάποια ζουμερά ερωτήματα για να απαντήσετε. Λοιπόν, ο πρώτος γύρος απαντήσεων. Έχουμε τέσσερα ακόμα μέλη που ετοιμάζονται να υποβάλουν ερωτήσεις. Παρακαλούμε λοιπόν να αφήστε κάποιο χρόνο για μετά, για τον επόμενο γύρο. Καλώς λέει ο κ. Παπαδήμος. Θα ακολουθήσει τη σειρά των ερωτήσεων, παρόλο που υπάρχουν συσχετισμοί μεταξύ των ερωτήσεων. Το πρώτο θέμα που τέθη είναι κα, ε, κατά πόσο εκτιλήσεται ακόμα η κρίση και τι κίνδυνοι υπάρχουν και αν οι κίνδυνοι συνεπάγονται και έναν δεύτερο γύρο τραπεζικής κρίσης. Εν γέννη δεν περιμένουμε να ισχύσει κάτι τέτοιο, παρόλο που είναι ξεκάθαρο ότι το τραπεζικό σύστημα στην Ευρωζώνη αλλά και γενικότερα στην Ένωση εξακολουθεί να προσαρμόζεται. Η διαδικασία μόχλευση συνεχίζεται, παρόλο που βλέπουμε ότι υπάρχει ύφε μείωση του ποσοστού, δεν αποκλείεται ότι το επόμενο έτος, σαν αποτέλεσμα της μέτριας οικονομικής δραστηριότητα, η απόλυση των δανείων ή οι χρεοκοπίες και μη αποπληρωμές των ε, δανείων θα συνεχιστούν και υπάρχει ο κίνδυνος να δημιουργηθεί ανάδραση και να επηρεαστεί η πραγματική οικονομία και ο τραπεζικός τομέας και το χρηματοστικό σύστημα. Και η αβεβαιότητα και η κίνδυνη όσον αφορά τη βιωσιμότητα του οικονομικού συστήματος αυξάνουν την αβεβαιότητα τη γενικότερη και αυξάνουν τον κίνδυνο, του κινδύνους που αντιμετωπίζει το τραπεζικό σύστημα. Εν γέννη όμως, νομίζω ότι έχουμε εξέλθει από την κρίση του τραπεζικού συστήματος και η αναμενόμενη ανάκαμψη της οικονομίας, αν και μέτρια, θα βοηθήσει την υποστήριξη των θετικών εξελίξεων. προτάθηκε και αναφέρθηκε ότι ένα πρόγραμμα οικονομικής σφαιρικής προσέγγισης που θέλει να μειώσει τα δημοσιονομικά ελλείμματα από πολύ ψηλά επίπεδα στο κάτω από τα 3% συνεπάγεται σοβαρή οικονομική ύφεση. Και ποιες είναι οι συνέπειες αυτού. Θα έλεγα εν γέννη ότι δεν θα πρέπει αυτομάτως να συμπεραίνουμε ότι αυτή η οικονομική προσέγγιση επί σειρά ετών τα οικονομικά μέτρα θα έχουν αντίθετα αρνητικά αποτελέσματα όσον αφορά την οικονομική ανάπτυξη, και οικονομικές επιδόσεις. Εγώ θα έλεγα το αντίθετο μάλιστα. Και είναι σημαντικό να κάνουμε διάκριση μεταξύ βραχυπρόθεσμων προσωρινών συνεπειών, που ίσως να είναι αρνητικές, αυτής της προσέγγιση οικονομική τη ενοποιημένη με μακροπρόθεσμα θετικά αποτελέσματα όσον αφορά την οικονομική δραστηριότητα που θα πρέπει να αναμένονται αυτά τα αποτελέσματα και πράγματι για αυτό το λόγο αυτή η ενοποίηση οικονομική και φορολογική και η βιωσιμότητα των δημοσιονομικών θεωρούνται στόχοι θεμελιώδης οικονομική. Αν δεν ληφθούν αυτά τα μέτρα, τότε αναπόφευκτα ο αντίκτυπος στα επιτόκια και η επιρροή στον ιδιωτικό τομέα θα δημιουργήσουν αρνητικά αποτελέσματα όσον αφορά την οικονομική δραστηριότητα στον ιδιωτικό τομέα. Στόχος των υγιών δημοσιονομικών και των βιώσιμων φορολογικών οικονομικών είναι υποστήριξη της οικονομικής ανάπτυξης μακροπρόθεσμα. Και περιμένω ότι σε χώρες που κάνουν δέουσες οικονομικές φορολογικές προσαρμογές βραχυπρόθεσμα, ότι οι χώρες αυτές θα ωφεληθούν μακροπρόθεσμα. Θα ωφεληθούν από τις συνέπειες αυτών των προσαρμογών λόγω του χαμηλότερου κόστους χρηματοδοτήσεω στο τέλο και τη απελευθερώσεως πόρων που θα είναι διαθέσιμη για την υποστήριξη τη ιδιωτική οικονομία. Και θα προσέθετα επίση ότι εφόσον, όσο προχωρούν αυτά τα οικονομικά μέτρα, η εμπιστοσύνη που επηρεάστηκε αρνητικά στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες θα αποκατασταθεί. Και αν ταυτόχρονα, και τώρα έρχομαι στο τρίτο ερώτημα που θέσατε, αυτέ οι προσαρμογέ οικονομικέ και φορολογικές συνδυαστούν με δομικές μεταρρυθμίσεις που βελτιώνουν την παραγωγικότητα στην οικονομία και βελτιώνουν τη διεθνή ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, αυτή είναι, αυτός είναι άλλος ένας διάβλος μέσω του οποίου οι οικονομικές δραστηριότητες στηρίζονται. Εγώ συμφωνώ ότι τα τελευταία χρόνια η οικονομική υποπτία και ο έλεγχος στην Ευρωζώνη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση εν γέννη δεν ήταν επαρκή για την, δημοσιο... για την αναγκαία οικονομική φορολογική πειθαρχία κατά τη διάρκεια της καλής εποχής οικονομίας, διότι την καλή εποχή πρέπει να δημιουργηθούν αυτοί, αυτοί τα φορολογικά, αν θέλετε, αυτά τα, αυτά τα αποθέματα για να απαλύνουν τα αποτελέσματα της κρίσης και, τα, και δεν ήταν και αποτελεσματικός ο έλεγχος. Ο έλεγχος έγινε αλλά δεν έγινε σωστή αξιολόγηση ίσως του αντιχτύπου της αυξήσεως αποκλήσεων ανταγωνιστικών και οικονομικών ανισορροπιών που επηρεάζουν τις οικονομίες των χωρών που υποφέρουν από τη μείωση ανταγωνιστικότητας αλλά και επηρεάζουν και τη συνοχή των οικονομίων της Ευρωζώνης. Τώρα βλέποντας προς το μέλλον και το ανέφερα αυτό ο στην εισαγωγή μου. Λοιπόν, βλέποντας το μέλλον τι θα γίνει. Προσβλέπουμε σε, κάποια πράγματα. Πρώτα απ' όλα θα ενισχυθεί, πιστεύουμε, το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης στο θεσμικό πλαίσιο εκείνο που θα βοηθήσει να αποφευχθεί η σώρευση οικονομικών ανισορροπιών και την εφαρμογή θετικών δράσεων εγκαίρως και συγχρόνως τη διεύρυνση της οικονομικής εποπτείας, ούτως ώστε να παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυς τις εξελίξεις τι αποκλίνουσες εξελίξει στη διεθνή ανταγωνιστικότητα και να προωθήσουμε τι αναγκαίε δράσει για την αποκατάσταση τη ανταγωνιστικότητα και τη βελτίωση τη αποδοτικότητα και τη συνοχή των οικονομιών τη Ευρωζώνης. Και πιστεύω ότι η νέα Task Force θα υποβάλει σχετικώ προτάσει. Τώρα σχετικά με το ρόλο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στις διαπραγματεύσεις, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι εταίρος κυρίως βασικά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Εθνές Νομισματικό Ταμείο και θα συμβάλλει η ΕΚΤ στην προετοιμασία του προγράμματος μαζί με τις ελληνικές αρχές και αυτή η προσπάθεια θα πρέπει να ολοκληρωθεί πριν ληφθεί η αδίποτε απόφαση όσον αφορά την εργοποίηση του μηχανισμού στήριξης και βεβαίως η δική μας συμβολή θα τονίσει ιδιαίτερα θέματα που σχετίζονται με τι διάφορε οικονομικέ προσαρμογέ που στο επίκεντρο του προγράμματος, αλλά, και πιστεύω στην προηγούμενη ερώτηση, και επί των μεταρρυθμίσεων που θα βοηθήσουν να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα τη ελληνική οικονομία Και ίσω κάτι γενικό το οποίο θα ήθελα να αναφέρω και να τονίσω και να υπογραμμίσω και το τόνισε επανειλημμένα και η Πρόεδρος. Είναι πολύ σημαντικό, πιστεύω, στις οικονομίες τη Ευρωζώνης οι εθνικέ οικονομικέ πολιτικέ και οι φορολογικέ και και οι διαθωτικέ αλλαγές και οι πολιτικές για την αγορά εργασίας να σχεδιάζονται και να εφαρμόζονται ούτω ώστε να συνάδουν με το στόχο της ΕΚΤ και της ενιαίας νομισματικής πολιτικής να παραμείνει ο πληθωρισμός κοντά και κάτω το 2%. 2%. Είναι θεμελιώδες αυτό το νούμερο για το σχεδιασμό και εφαρμογή των εθνικών οικονομικών πολιτικών διότι δεν γίνεται μακροπρόθεσμα τα, οι εθνικοί πληθωρισμοί συστηματικά επίμονα να αποκλίνουν σημαντικά από το 2%. Και αυτό μπορεί να είναι ένα σημείο που να καθορίζει φορολογική πολιτική ε, και πολιτική στην αγορά εργασία και οικονομική πολιτική. Η πρακτική συμμετοχή της ΕΚΤ σχετίζεται μόνο με το ρόλο φορέα διευκόλυνσης των πληρωμών, αλλά δεν θα παρά, δεν θα δώσουμε χρήματα σαν έκτεν, έχουμε άλλο ρόλο να παίξουμε σε αυτό. Ναι, έχουμε και χρονικούς περιορισμούς, άρα έχουμε μια κρίση χρονική. Για τις πιέσεις στην αγορά υπήρξαν διάφοροι παράγοντες που επηρέασαν την αντίδραση της αγοράς, κυρίως ανησυχίες για την οικονομική βιωσιμότητα της Ελλάδας και τη δυνατότητα που έχει η χώρα να αναχρηματοδοτήσει το χρέος της σε βραχυπρόθεσμα. Υπάρχουν και άλλες αβεβαιότητες και παράγοντες που έπαιξαν ρόλο, αλλά αυτό που είναι σημαντικό τώρα είναι να δούμε στο μέλλον και να δούμε πώς αυτό το πρόγραμμα το οποίο ετοιμάστηκε μπορεί να ολοκληρωθεί και να εφαρμοστεί επιτυχώς και εγκαίρως. Τώρα όσον αφορά το άλλο που αναφέρθηκε για το ότι υπογραμμίζει συχνά η ΕΚΤ τις δαπάνες για την μείωση των ελλημάτων. Να πω δύο πράγματα εντάχει. Πρώτα απ' όλα συμφωνώ ότι το μέγεθος του δημοσίου τομέα απαραίτητα δεν αποτελεί δείκτη της αποδοτικότητας του τομέα, όμως συχνά είναι. Όχι απαραίτητα, συχνά. Αν δούμε λοιπόν την εμπειρία που έχουμε από διάφορε χώρε επί σειρά ετών, παρόλο που συμφωνώ ότι δεν είναι αυτομάτω κάτι που ισχύει και υπάρχουν παραδείγματα χωρών που έχουν συνδυάσει σχετικά μεγάλο δημόσιο τομέα με αποδοτικό τέτοιο δημόσιο τομέα, σε άλλε περιπτώσει σε πολλές άλλες περιπτώσεις έχουμε πολύ κακές εμπειρίες και αυτό που θέλουμε να πούμε δεν είναι κάτι πολιτικής φύσεως, διότι είπα αυτό ακριβώς τα εισαγωγικά μου σχόλια. Είπα ότι εστιαζόμενοι στις δαπάνες αυτό είναι σημαντικό, διότι η εμπειρία έχει καταδείξει ότι είναι αποτελεσματικότερο τρόπο βάσει των στοιχείων που έχουμε στη διάθεσή μα, με τον οποίο μπορούμε να πετύχουμε πλέον μόνιμη και βιώσιμη μείωση των οικονομικών ανισορροπιών. Αν αυτό μπορεί να επιτευχθεί διαφορετικά, βεβαίω αυτό είναι ευθύνη των οικονομικών αρχών, αλλά να φέρουμε την εμπειρία η οποία μας έδωσε τα αποτελέσματα. Δεν τα δεν το ερμηνεύω αυτό. Δεν είναι πολιτική δήλωση, απλώς είναι μια δήλωση που σχετίζεται με την όλη ιστορία και τα στοιχεία που έχουμε συλλέξει. Ευχαριστώ. Έχουμε όπως πάντα πρόβλημα χρόνου <clears throat> γιατί θέτουμε ερωτήματα τα οποία απαιτούν λεπτομεριακές απαντήσεις. Έχουμε έξι ακόμα ομιλητέ που θέλουν να λάβουν το λόγο. Κανένα άλλο δεν θα λάβει το λόγο. Θα ακούσουμε και του έξι μαζί. Θεωρητικά έχουμε τέσσερα λεπτά ακόμα, αλλά θα ξεπεράσουμε λιγάκι κατά 15 λεπτά το, το χρόνο που προβλέπαμε, γιατί δεν ξεκινήσαμε εγκαίρως, ξεκινήσαμε ένα θέατρο καθυστέρηση. Παρακαλώ ένα, ερωτήματα, ένα ερώτημα θέλ, να θέσετε και να παραμείνετε στα πλαίσια ενός λεπτού. Ο κύριος Χούντης έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Παπαδήμα, κύριε Αντιπρόεδρε, χαίρομαι που σας είστε εδώ και σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας και για την παρουσίαση που κάνατε. Το ερώτημα που θα σας κάνω έχει σχέση προφανώς με τα θέματα που εξελίσσονται σήμερα στην Ελλάδα, αλλά η απάντησή σας προφανώς δεν θα είναι απάντηση ως Έλληνα, αλλά ως ε, ε, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Το πρώτο ερώτημα τι αισθήματα σας δημιουργεί στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα η για πρώτη φορά συμμετοχή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου σε υποθέσεις της Ευρωζώνης. Γιατί ήταν απαραίτητη αυτή η συμμετοχή. Εν πάση περιπτώσει δεν πήρατε εσείς την απόφαση. Τι συμπεράσματα βγάζετε. Έχετε ανησυχίες, συμφωνείτε. Λέω η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα βλέπει κάτι ε, πιο δραματικό στην περίπτωση που αυτός ο μηχανισμός ενεργοποιηθεί αύριο για την Πορτογαλία και για την Ισπανία. Και το δεύτερο ερώτημα συμπληρωματικό. Στην πρώτη περίπτωση ναι, είναι η θεσμική, δεν προβλεπόταν από πουθενά αυτή η συνθήκη. Αλλά πρακτικά, πρακτικά αν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο υποβάλει καινούριου όρους ενώ εσείς έχετε και είναι ικανοποιητικό το πρόγραμμα δημοσιονομικής εξυγίανσης. Ποιος θα είναι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σε μια τέτοια διαφωνία. Ευχαριστώ, Σβέν. Σα παρακαλώ και πάλι μου, συνάδελφοι, να είμαστε σύντομοι, γιατί αλλιώ δεν θα απαντήσει ο, ο κύριο Αντιπρόεδρο. Δεν είναι δίκαιο για τον κύριο Παπαδήμο να τον αφήσουμε μονάχα με τρία λεπτά για να απαντήσει 20 ερωτήματα. Ο Σβέν Γκίκολτ έχει το λόγο. Πάρα πολύ σύντομα. Διαβάζοντα την ετήσια έκθεσή σα τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, θέλω να υπογραμμίσω ότι το θέμα των εσωτερικών ελλείψεων ισορροπίας και οι αποκλήσει μεταξύ κρατών μελών δεν αντανακλώνται πλήρω κατά τη δική μου άποψη στην έκθεση αυτή. Αντιμετωπίζονται σωστά όταν πρόκειται για τα δημόσια οικονομικά, αλλά όταν πρόκειται για την νομισματική πολιτική και τα αποτελέσματα τη νομισματική πολιτική, η έκθεση νομίζω ότι είναι κάπω αποδυναμωμένη. Επιπλέον, δεν θέλω να θέσω ένα ερώτημα, απλώ θέλω να κάνω μια παρατήρηση μετά από την επίσκεψη που κάναμε στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ανησυχούμε πάρα πολύ για τα εργασιακά δικαιώματα στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και θεωρούμε ότι πρέπει να ακολουθήσετε τα διεθνή πρότυπα για το πώς αντιμετωπίζετε τα συνδικάτα στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Υπάρχουν πολλά που πρέπει να γίνουν και περιορίζω μονάχα σε αυτό το επίπεδο. Για να μείνουμε στο χρόνο μου. <clears throat> Ευχαριστώ. Η Κάθριν έχει το λόγο. Η Κάθριν Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ τον κύριο Παπαδήμο επίσης. Ένα σύντομο ερώτημα σε σχέση με τα κύρια διδάγματα τα οποία μπορούμε να αντλήσουμε από την ελληνική κρίση. Αν δω την έκθεσή σας της Κεντρικής Τράπεζας και αυτά που λένε οι σχολιαστές, λένε πάρα πολύ ότι και η Πορτογαλία είναι σε μια δύσκολη κατάσταση. Λέει η έκθεσή σας την. Ε, ότι η Πορτογαλία βρίσκεται σε μεγάλο κίνδυνο σε ό,τι αφορά τη βιωσιμότητα των ε, <clears throat> οικονομικών της. Ενώ χώρες όπως το Βέλγιο, Ιταλία, Γερμανία, Λουξεμβούργο, Αυστρία και Ιταλία βρίσκονται σε μεσαίο κίνδυνο. Ανησυχώ λοιπόν, αν δεν μάθουμε τα διδάγματα από την ελληνική κρίση, τι θα γίνει, τι θα μπορούσε να γίνει στο μέλλον με όλες αυτές τις χώρες. Και τέλος, Ποιο θα σας αντικαταστήσει στο αξίωμα του Αντιπρόεδρου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας. Η Επιτροπή μας έχει εγκρίνει ήδη την αντικατάσταση του κύριου Παπαδήμου. Θα είναι ο κύριος Βίκτορ Κωνστάνσιου, ο αντικαταστάτης του κύριου ε, Παπαδήμου. Ο κύριος ε, Ούντο Μπούλμαν έχει τώρα το λόγο. Κύριε Παπαδήμο, εξ ονόματος σοσιαλιστικής ε, ομάδος, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα τελευταία χρόνια, για την παρουσία σας, για τον τρόπο με τον οποίο είχατε διατηρήσει μια πολύ καλή επικοινωνία με την Επιτροπή μας μέσα σε δύσκολες κατάστασεις, όχι μονάχα δύσκολες καταστάσεις για την Ελλάδα και για άλλες χώρες. Η Κομισιόν ανέφερε το ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ευρωπαϊκούς μηχανισμούς και αναφέρθηκε ακόμα και ένα ευρωπαϊκό ταμείο, μια διευκόλυνση για τα θέματα αυτά. Πώ θα εξασφαλίσουμε όμω ότι στο μέλλον δεν θα υπάρχουν κερδοσκοπικέ κινήσει κατά των κρατών μελών τη Ευρωπαϊκή Ένωση, Κύριε Παπαδήμου, θα ήθελα να ξέρω ποια είναι η άποψή σα σε σχέση με την πρόταση δημιουργία ενό Ευρωπαϊκού Ταμείου και εφόσον είναι και η τελευταία σας εμφάνιση ενώπιόν μα, εγώ δεν θα είχα κανένα πρόβλημα να μιλήσετε ειλικρινά σε εμά και όχι απλώ να αναφέρετε την επίσημη θέση τη ΕΚΤ. Εντάξει, <clears throat> τελευταίοι δύο μιλητές, ο Βέρνερ Λάγκεν και Άννη Λίγκεν. Βέρνερ, όχι, δεν θέλεις να λάβεις το λόγο. Γιάννη και, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Έχω να σας θέσω δύο ερωτήματα. Καταρχήν, μεταρρύθμιση αυτή για την... Ε, δεν έχουμε μετάφραση, λέει πρόεδρος. Μια στιγμή, <clears throat> μην, μην προχωρείτε τόσο γρήγορα. Το πρώτο μου ερώτημα έχει να κάνει με την μεταρρύθμιση της εποπτείας. Είπατε ότι είναι πολύ σημαντικό να αλλάξει το σύστημα μακροπολιτικής εποπτείας και ότι θα έχουμε ένα νέο σύστημα το οποίο θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2011. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μιλάμε όλο και περισσότερο για μια ευρωπαϊκή λύση σε ό,τι αφορά τις τράπεζες οι οποίες έχουν διασυνοριακό χαρακτήρα και θέλουμε να θεσπίσουμε ένα ευρωπαϊκό σύστημα εποπτείας για αυτές τις τράπεζες. <clears throat> Στο Συμβούλιο Κοφίν υπήρξε μια πρόταση σχετικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρόκειται λοιπόν για... Αλλά αυτό το οποίο προτάθηκε εκεί ήταν εθνικοί ρυθμιστές με ευρωπαϊκά στοιχεία συντονισμού. Δεν είναι αρκετά φιλόδοξο το Συμβούλιο κατά την άποψη του Κοινοβουλίου που θέλει η Ευρωπαϊκή Αρχή. Ποια είναι η άποψή σας σχετικά. Ένα δεύτερο ερώτημα το, η Ειδικούσα Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου φαίνεται ότι δεν θα εκπροσωπηθεί η Eurostat. Ποια είναι η απόψή σας σχετικά. Εντάξει, όσο πιο σύντομα μπορείτε κύριε Παπαδήμου. With regard to the involvement, uh, Όσον αφορά τη συμμετοχή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, πάντα θα συμμετείχε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο όσον αφορά την παροχή τεχνογνωσίας και υποστήριξης. Ελήφθη απόφαση σε περίπτωση ενεργοποίησης του μηχανισμού στήριξης οι χώρες της Ευρωζώνης και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θα συμβάλλουν ταυτόχρονα. Πιστεύουμε ότι είναι εφικτή λύση και αυτό που είναι σημαντικό είναι το πρόγραμμα το οποίο ετοιμάζεται, όπως προανέφερα, να ολοκληρωθεί εγκαίρως και να ασχοληθεί με τα αίτια των οικονομικών και διαθετικών προβλημάτων της Ελλάδας. Πιστεύω ότι θα υπάρξουν δυσκολίες όσον αφορά κοινή θέση, ίσως και διαφορές θα υπάρξουν κατά τις διαπραγματεύσεις, θα επιληθούν και θα επιτευχθεί συμφωνία. Όλοι οι θεσμοί που συμμετέχουν και η ελληνική κυβέρνηση έχουν κοινούς στόχους. Πιστεύω ότι η έκθεσή μας τονίζει επαρκώς τις εσωτερικές ανισορροπίες της Ευρωζώνης και στις παρουσιάσεις και τις ακροάσεις του Προέδρου και σε άλλα βήματα συζητήσεων τονίζεται η σημασία στενής παρακολουθήσεως των ισορροπιών και διαφορών ανταγωνιστικότητας συστηματικά υπογραμμίσαμε επί σειρά ετών αυτό το θέμα. Όσον αφορά τα συνδικάτα, τα τελευταία χρόνια η θέση των συνδικάτων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ενισχύθηκαν. Αναγνωρίσαμε, ως γνωρίζετε, ε, τα συνδικάτα και το ρόλο τους πρόσφατα. Τα βασικά μαθήματα από την οικονομική κρίση της Ελλάδας τα μάθαμε, πιστεύω. Τα μάθαν πρώτα απ' όλα στην Ελλάδα και οι αρχές και ο λαός καταλαβαίνουν την ανάγκη που υπάρχει να επιτευχθούν οι στόχοι, δηλαδή να ακολουθηθούν θέσεις οικονομικές υγιής και να γίνουν και μεταρρυθμίσεις αναγκαίες για να είναι πιο αποδοτική οικονομία. Παρόμοια προβλήματα σε διαφορετικό βαθμό αντιμετωπίζονται από άλλες χώρες. Κάποιες χώρες έχουν περισσότερη δουλειά να κάνουν όσον αφορά την οικονομική πολιτική, Άλλες χώρες πρέπει να προχωρήσουν πολύ στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητά τους. Τα πρόσφατα γεγονότα ήταν ένα συναγερμός αν θέλετε, μας ξύπνησε αυτό για να προσαρμόσουμε τις πολιτικές δεόντως, για να αποκαταστήσουμε την ανταγωνιστικότητα και να πετύχουμε σωστή οικονομική τοποθέτηση. Μπορεί να πει κανείς ότι αυτά είναι τα θετικά αποτελέσματα, ο αντίκτυπος ο θετικός της ελληνικής κρίσης επί άλλων οικονομιών που αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα. Το ευρωπαϊκό μέσο στήριξης που περιγράψατε είναι μεγάλο πρόγραμμα, έχει πολλές προκλήσεις, ε, το θέμα είναι πώς θα καθοριστεί και θα είναι τα χαρακτηριστικά. Η προσωπική μου άποψη και της τράπεζας είναι ότι πρωτίστως στο άμεσο μέλλον πρέπει να ενισχύσουμε το θεσμικό πλαίσιο που υπάρχει και να το συμπληρώσουμε. Να ενισχύσουμε το Σύμφωνο Σταθερότητα και Ανάπτυξη, αλλά να συμπληρώσουμε και την εποπτεία και μέσω τη διευρύνσεω και τη ενισχύσεω εποπτεία να αποφύγουμε νέε κρίσει. Η πρόληψη, πιστεύω, πρέπει να τονιστεί. Καλύτερη πρόληψη, καλύτερα τονιστεί η πρόληψη παρά μηχανισμοί που μπορούν να βοηθήσουν να αντιμετωπιστεί μια κρίση όταν συμβεί. Τώρα, ο ακριβής μηχανισμός που θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί απαιτεί προσεκτική ανάλυση και προβληματισμό, διότι θα πρέπει να συνάδει με τις διατάξεις των συνθήκων και πιο συγκεκριμένα με τις διατάξεις για την μη οικονομική ενίσχυση για να γλιτώσει μια οικονομία και θα πρέπει να αντιμετωπιστούν τα διάφορα συναφή προβλήματα να ακολουθηθεί σωστή διδολογική προσέγγιση. Τα μέτρα θα πρέπει να αντιμετωπίζουν την κρίση και ταυτόχρονα θα πρέπει να, να ενισχύονται οι προσαρμογές για την αποφυγή επανάληψης, μελλοντικής επανάληψης κρίσης. Και τώρα τα δύο άλλα θέματα που εφήγησαν για την εποπτική μεταρρύθμιση. Εκτιμούμε τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής σας. Πιστεύουμε όμως ότι οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αφορούν τον πυλώνα της ε, μικροοικονομικής συνετής διαχείρισης πιστεύουμε ότι οι εθνικές αρχές φέρουν την ευθύνη τη βασική για την καθημερινή εποπτεία και τον έλεγχο. Όμως μεταρρύθμιση χρειάζεται στον τομέα αυτό που συνεπάγεται ενίσχυση συντονισμού και συνεργασίας στο μικροοικονομικό τομέα για τη συνετή διαχείριση και στη διαχείριση της οικονομίας και για να αντιμετωπιστούν μελλοντικές ε, παρόμοιες κρίσεις. Ε, ευχαριστώ για την υπομονή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα μπορούσαμε να σας κρατήσουμε εδώ ε, για όλη την πρωινή μας συνεδρίαση. Δυστυχώς όμως έχουμε πολλά πράγματα να συζητήσουμε, καθώς και το πακέτο εποπτείας και άλλα θέματα. Αλλά εφόσον είναι η τελευταία φορά που ήρθατε εδώ, σας ευχαριστώ εκ νέου για τις προσπάθειές σας που κάνατε αυτά τα χρόνια και για τον τρόπο με τον οποίο προσπαθήσατε πάντα να απαντήσετε σε ερωτήσεις μας. Και μάλιστα σε έναν πολύ σύντομο χρόνο που σας διαθέτουμε και είναι άδικο για σας. Ευχαριστούμε. Σας ευχόμεθα ό,τι καλύτερο για το μέλλον. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο κ. Παπαδήμος. Εκτιμώ το ότι είχα την ευκαιρία να εμφανιστώ μπροστά σας και να συμμετάσχω στη συζήτηση. Αγαπητοί συνάδελφοι, πάμε στις ψηφοφορίες σε δύο λεφτά. Σας δίνω μερικά δευτερόλεπτα για να αυτοοργανωθείτε με τους καταλόγους ψηφοφορίας. Και να μπορέσω να αποχαιρετήσω τον καλεσμένο μας. Ελπίζω ότι έχετε τις κάρτες σας, όχι τις πιστοτικές, αλλά τις κάρτες ψηφοφορίας, αγαπητοί συνάδελφοι, για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε. Αγαπητά μέλη, μήπως μπορούμε να ξεκινήσουμε. Νομίζω ότι αυτά τα θέματα δεν είναι ιδιαίτερα αμφιλογόμενα. Ανοίγουν και τα παράθυρα για αυτούς που θέλουν λίγο φως, τα ρολά μάλλον ανεβαίνουν για αυτούς που θέλουν φως τα είχαμε κατεβάσει γιατί υπήρχε βιδεοσκόπηση της ε, παρουσίας του Αντιπρόεδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και χρειαζόταν ειδικό φωτισμός. Αλλά τώρα μπορούμε να ρίξουμε άπλετο φως στη δημοκρατική διαδικασία ψηφοφορίας. Ξεκινάμε με την πρώτη ψηφοφορία, σημείο 10 της ημέρας διάταξης, ο κανονισμός για τη συνολική εξαίρεση αυτοκίνητων οχημάτων και από ό,τι μου λένε δεν υπάρχει αντίρρηση να ψηφίσουμε όλο το κείμενο από κοινού. Μπορούμε να ψηφίσουμε λοιπόν το αρχικό κείμενο όλο ομού. Όλοι αυτοί που είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. Το κείμενο όπως έχει τροποποιηθεί ψήφι κατά αποχές εγκρίνεται. Σημείο 11. Το σχέδιο ψηφίσματος τώρα για τον κανονισμό συνολικών εξαιρέσεων στον τομέα των αυτοκινήτων οχημάτων. Έχουμε κάποιες συμβαστικές τροπολογίες. Ελπίζω ότι δεν θα είναι πολύ δύσκολη ψηφοφορία. Πρώτη τροπολογία, τροπολογία 1 των σοσιαλιστών Ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στη συμβαστική τροπολογία 1. Α μάλλον ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ψήφισμα την παράγραφο 3, το αρχικό κείμενο, υπέρ, κατά, εποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 4 των σοσιαλιστών κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία Β, ψήφι υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία C, ναι, Παράγραφος 6, αρχικό κείμενο. <clears throat> ναι. Παράγραφος 6, αρχικό κείμενο. Πρέπει να την ψηφίσουμε. Εφόσον χρειάζεται να την ψηφίσουμε. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τώρα συμβαστική τροπολογία C. Ναι, είναι λιγάκι πολύ σκιερά και σκιασμένα όλα αυτά. Τροπολογία 6β του ΕΛΚ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τώρα επιτέλους πάμε στη συμβαστική σε ψήφι περ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική D, ψήφι περ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική ή λατινικό τμήμα α ψήφι υπέρ. Εντάξει. Συμβαστική ή τμήμα α. Σύμφωνοι. Ψήφι υπέρ. Κατά. Ας ελέγξουμε λοιπόν ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέραν της κυρίας Λούλινγκ. Ποιος άλλος έχει δυσκολία να ψηφίσει ηλεκτρονικά. Έχουμε ξεκινήσει. Πρέπει να ξαναψηφίσουμε. Άρχεται και πάλι ψηφοφορία. Πέρας. Αν δεν δουλεύει το μηχάνημά σας, πηγαίνετε, πηγαίνετε δίπλα στην επόμενη πέρας προφορία λοιπόν, πέρας. Μα τι έχετε πάλι, τι πάθατε πάλι. Έχουμε πολλούς σοσιαλιστές, παραπάνω από τον κανονικό αριθμό που ψηφίζουμε, λέει η πρόεδρος. Τώρα είναι εντάξει. Δεν μπορούμε να είμαστε πάρα πολλοί. Είμαστε όσοι πρέπει, λέει κάποιος από τους σοσιαλιστές στις προφορίες. Απορρίπτεται λοιπόν η τροπολογία αυτή. Συμβαστική ε τμήμα β. Ψήφι υπέρ παρακαλώ. Γιατί δεν ψηφίζετε. Σηκώστε τα χέρια σας όχι μόνο οι συντονιστές και τα μέλη να ψηφίζουν ψήφι κατά αποχές. Νομίζω ότι εγκρίνεται. Συμβιβαστική. Θέλετε πράγματι να ελέγξουμε. Όχι. Τότε γιατί το ζητάτε. Συμβιβαστική ε τμήμα C. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 7 δέλτα. Ψήφι υπέρ παρακαλώ. Τροπολογία του ΕΛΚ. Ίσως θέλετε να ψηφίσετε υπέρ του κόμματός σας. Λοιπόν, ψήφι υπέρ. Πρέπει να μετρήσω και τα χέρια σας. Άμα δεν τα σηκώσετε δεν σας μετρήσω. Ζων Πολ, μπορείς να μαζέψεις τα πρόβατά σου, να μαζέψεις την ομάδα σου, να ψηφίσεις. για την 7 Δέλτα. Ψήφι υπέρ. Ψήφι υπέρ λοιπόν. Κατά. Αποχές δεκτή. Συμβαστική F σίγμα δηλαδή τμήμα α, ψήφι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική F τμήμα β ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 8 της ΓΟΕ, ψήφι υπέρ, κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική G, ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική H, λατινικό τμήμα α, ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Συμβαστική H, τμήμα β, ψήφι υπέρ. Έχουμε χωριστή ψηφοφορία εδώ που έχει ζητηθεί από το... Έχουμε τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα, κατά αποχές νομίζω ότι εγκρίνεται αλλά πρέπει να το ελέγξουμε μάλλον πρώτο τμήμα της συμβαστικής H τμήμα Β πέρας ελπίζω εγκρίνεται Δεύτερο τμήμα τώρα. Ψήφι υπέρ. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Το δεύτερο τμήμα του πρώτου τμήματος είναι λιγάκι μπερδευτικά. Ψήφι υπέρ, εν πάση περιπτώσει. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται με την διαπλειοψηφία τρίτο κομμάτι του πρώτου τμήματος, αν θέλετε να ελέγξουμε. Λοιπόν, κάνουμε ψηφοφορία ελέγχου για το δεύτερο τμήμα του πρώτου τμήματος. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Με μεγαλύτερη πλειοψηφία εγκρίνεται. Τώρα ψηφίζουμε το τρίτο τμήμα, ψήφι υπέρ. Το τρίτο τμήμα του πρώτου τμήματος, ψήφι κατά, αποχές. Νομίζω ότι και εδώ υπάρχει έγκριση, αλλά θα κάνουμε έλεγχο. Άρχεται ηλεκτρονικός έλεγχος. Ψήφισατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική I, λατινικό ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Εννέα C, ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 9D ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβαστική J, ψήφι υπέρ. Τμήμα Α, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική J, τμήμα Β, όχι. Το τμήμα Β, Β εκπίπτει τη συμβαστική J. Σημείο 12, τροπολογία 12 μάλλον από τους σοσιαλιστές, ψήφι υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Παράφος 13. Ψήφι περ Κατά. Θα ψηφίσουμε μετά τις αιτιολογικές σκέψεις όλες μαζί. Αλλά την παράγραφο 13 πρέπει να ψηφίσουμε, ψηφίσουμε χωριστά. Παρακαλώ σηκώστε τα χέρια σας. Κατά. Απόχες. Εγκρίνεται. Μπορούμε να κάνουμε όλες τις αιτιολογικές σκέψεις, τροπολογίες από κοινού. Συμφωνείτε. Όλες οι αιτιολογικές σκέψεις μαζί, ψήφι κατά, αποχές, όλες εγκρίνονται. Περάσαμε τι αιτιολογικέ αναφορές. Είμαστε αιτιολογική σκέψη α του ΕΛΚ. Ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Αρχική αιτιολογική σκέψη α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη β υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Νέα αιτιολογική σκέψη σ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Εκπίπτει αρχική. Δέλτα υπέρ αρχική κατά αποχές. λογική ε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Αιτιολογική F υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Αιτιολογική G υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Νέα αιτιολογική H από το Elk. ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική K ψήφι υπέρ, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Αιτιολογική J, η αρχική υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Αιτιολογική K, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Νέα αιτιολογική σκέψη L από το ΕΛΚ, ψήφι υπέρ, Jean-Paul, το υποστηρίζεις κατά αποχές εγκρίνεται. Είναι συμβατή αυτή η αιτιολογική σκέψη με την ΕΛ των σοσιαλιστών. Ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. L α από το ΕΛΚ, ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. ΕΛ β από το ΕΛΚ υπέρ κατά αποχές Μήπω μπορούμε να ελέγξουμε, δεν κατάλαβα ακριβώ τι έγινε. LB, νέο. Από το κόμμα των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών είναι λίγο μπερδεμένα όλα αυτά τα πράγματα όπω καταλαβαίνετε, αλλά νομίζω ότι καταλαβαίνω τι γίνεται. Ψήφισατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη M από την ΚΟΕ, e, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. M αιτιολογική από τη σοσιαλιστική ομάδα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και νέα αιτιολογική σκέψη MA από το ΕΛΚ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τα έχουμε ψηφίσει όλα. Ωραία. Τελική ψηφοφορία στο κείμενο όπως έχει τροποποιηθεί. Ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια σε κάποιον. Εργάζεται και πολύ σκληρά ε, ε, και εργάζεται πολύ σκληρά η γραμματεία για όλα αυτά. Πάμε για το σημείο 12, για ε, την ψηφοφορία για το σημείο 12. Πρέπει να διαβάσω τις σημειώσεις της Προέδρου εδώ μου λέγουν. Υπάρχει ενδεχόμενη αναβολή του θέματος αυτού στην Ολομέλεια. Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στις 22 Απριλίου να αναβάλει απόφαση για τα επόμενα βήματα για τις γενικές κατευθυντικές γραμμές για την οικονομική πολιτική και την απασχόληση. Ο λόγος για την απόφαση της διασκέψεως των Προέδρων είναι ότι θεωρούμε ότι το Συμβούλιο δεν δίνει στο Κοινοβούλιο αρκετό χρόνο να αντιδράσει και αυτό αφορά ιδιαίτερα την Επιτροπή Απασχόλησης που υπέχει υποχρέωση να αναμένει τη γνωμοδότηση του Κοινοβουλίου αλλά επηρεάζει και μας. Θα συζητήσουμε αργότερα σήμερα στους συντονιστές το πώς μπορούμε να προχωρήσουμε, αν θα ψηφίσουμε την επόμενη εβδομάδα ή αν θα αποσταλεί επιστολή ή αν θα το κάνουμε μετά από την ανακοίνωση του Όλι Ρεν. Για την ώρα θα ασχοληθούμε το, με την προφορική ερώτηση. Δεν εξαφανίστηκε το σημείο από την ημερήσια διάταξη, αλλά υπήρξε το αίτημα της διασκέψεως των Προέδρων και πρέπει να δούμε που είμαστε, τι θέλουμε να κάνουμε και θα επιστρέψουμε. Προχωράμε και πάμε στη ψηφοφορία. Παράγραφος 1. Το αρχικό κείμενο. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ερώτημα 1 που υπευλήθη από το S&D υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ερώτηση 2. Υπευλήθη από το S&D υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Ερώτηση 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ερώτημα 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ερώτηση 5 όσα αναθεωρηθήκε από την άλλη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Αυτό είναι. Όλα τα άλλα έχουν καταπέσει. Ψηφίζουμε το τροποποιημένο κείμενο υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ όλους. Επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης είναι ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις τροπολογίες για το πακέτο το εποπτικό μας έχει δείξει εμπειρία κατά το παρελθόν ότι έχουμε πάρα πολλούς που θέλουν να μιλήσουν για το θέμα. Και δεν είμαι σίγουρη ότι θα έχουμε αρκετό χρόνο ούτω ώστε να μιλήσουν όλοι και να έχουμε δύο γύρους παρεμβάσεων από όλους τους εισηγητές. Παρακαλώ όλους λοιπόν να είναι σύντομοι και ας ξεκινήσουμε με μια σύντομη παρέμβαση κάθε εισηγητού που θα εστιάζεται στο που φτάσαμε όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις για συμβαστικές τροπολογίες. Υπενθυμίζω στα μέλη ότι θεωρητικά προσπαθούμε ακόμα να ψηφίσουμε. Well, have we got all the rapporteurs here that need to be here? Um, we are 10 minutes. Έχουμε προχωρήσει Έχουμε κερδίσει 10 λεπτά στο χρόνο μας, αλλά δεν θέλω να στερηθούμε αυτό το χρόνο τη συζήτηση, οπότε παρόλο που είμαστε μπροστά χρονικά, θα ήθελα να πάμε στο επόμενο θέμα. Είναι ενδεικτικό το χρονοδιάγραμμα, το ξέρετε όλοι. Να δώσω το λόγο καταρχάς στον εισηγητή της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής του Φορέα. Όσο πιο σύντομος είσαστε, τόσο περισσότερες πιθανότητες έχετε να μπορέσετε να δευτερολογήσετε. Θα είμαι σύντομος και όσο μπορώ πιο σαφής, λέει ο κύριος ε, Γκάρθια Μαργάλιο. Καταρχήν, σαν προκαταρκτικές παρατηρήσεις, οι κοινοβουλευτικές εργασίες είναι συλλογικές από την φύση τους, αλλά αυτή είναι ακόμα πιο συλλογική από τις συνηθισμένες ενέργειες, γιατί Καταρχήν βρισκόμαστε σε αχαρτογράφητες περιοχές και δεύτερον γιατί είναι απαραίτητο όλες αυτές οι εκθέσεις που έχουν να κάνουν με το πακέτο εποπτείας να διατρέχονται από μια κοινή φιλοσοφία. Θέλω να ευχαριστήσω λοιπόν τους συζητητές, τους κοιόδης συζητητές, όλους αυτούς οι οποίοι έχουν επίσης βοηθήσει στις διάφορες επιτροπές. Στην Συνταγματική Επιτροπή ενεκριθεί με η γνωμοδότηση με δύο μονάχα ε, αποχές. Είναι μια εργασία η οποία είναι συνεχιζόμενη. Σήμερα έχουμε μια συνεδρίαση με την οποία θα μπορέσουμε να συλλέξουμε τις απόψεις όλων των εισηγητών και συνεχίζουμε τις διαπραγματεύσεις πριν από την ψηφοφορία στην Επιτροπή μας και στη συνέχεια θα πρέπει να συνεχίσουμε πριν από την Ολομέλεια και μετά από την Ολομέλεια όταν θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε τις θέσεις του Συμβουλίου. Αυτό το οποίο θέλουμε τώρα είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μπορέσει να καταλήξει σε μια σταθερή και στεναρή θέση για τις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο που αυτή τη στιγμή είναι πολύ δύσκολο να ξέρουμε ποια θα είναι η πορεία της και τα αποτελέσματά της. <clears throat> Μετά από την εξέταση των τροπολογιών, εγώ έχω καταλήξει σε ένα ενοποιημένο κείμενο που περιλαμβάνει τις τροπολογίες που έχω δεχτεί και αυτές που δεν έχω δεχτεί ακόμα και αυτές που έχω δεχτεί μονάχα εν μέρη. Είναι μια προσωρινή εργασία που βέβαια θα συνεχίσει να τροποποιείται κατά τη διάρκεια της εξέτασης και νομίζω ότι θα προσπαθήσω να δίνω σε όλους τους βουλευτές τις ε, αλλαγές που γίνονται σε πραγματικό χρόνο για αυτή την έκθεση. Επίσης, στην κρίση των τροπολογιών εγώ έλαβα υπόψη τις προηγούμενες κοινοβουλευτικές εκθέσεις από το 2000 μέχρι πρόσφατα <clears throat> και συγκεκριμένα της Ελίζα Φερέιρα σε ό,τι αφορά τη διαχείριση της κρίσης. Εμείς ξεκινήσει όλοι οι συγητές και εγώ φυσικά από το κείμενο της Κομισιόν και όχι του Συμβουλίου. Το κείμενο του Συμβουλίου έχει εξεταστεί από τους συντονιστές των κύριων πολιτικών ομάδων λέγοντας ότι ήταν ένα κείμενο απαράδεκτο σε ό,τι αφορά το περιεχόμενό του. Η κοινοβουλευτική λοιπόν έκθεση που παρουσιάζω βασίζεται σε τρεις βασικές αρχές. Θεωρούμε ότι το θέμα που αντιμετωπίζουμε είναι θέμα εσωτερικής αγοράς. Πρέπει να σταματήσουμε την, τον κατακαιρματισμό σε επίπεδο κανόνων και την ανομοιογένεια τη εσωτερική αγορά. Είναι επίση απαραίτητο να έχουμε καλύτερη εποπτεία, είναι απαραίτητο να αποφύγουμε του κινδύνου για του φορολογούμενους για να μην υπάρξει στο μέλλον το κόστος μιας κρίσης που θα το επομιστεί το θυλάκιο του φορολογούμενου. <clears throat> Γι' αυτό δεν έχω λάβει υπόψη πολλές τροπολογίες που έχουν διατυπωθεί από πολλές ε, πολιτικές ομάδες, γιατί τονίζουμε ότι είναι οι δημόσιες αρχές οι οποίες θα πρέπει να εξασφαλίσουν την λειτουργία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, την προστασία των φορολογούμενων και των κύριο θεσμικών οργάνων. Πρέπει εμείς λοιπόν να προβούμε σε μια ε, καλύτερη ρύθμιση των αγορών και δεν μπορούμε να περιμένουμε ότι οι αγορές από μόνες τους θα αυτοοργανωθούν και θα αυτορυθμιστούν. Εκεί που υπάρχουν οι μεγαλύτερες διαφορές σε σχέση με το κείμενο της Κομισιόν και του Συμβουλίου, ξεκινώ με το θέμα των κανόνων. Το κείμενο της Κομισιόν μιλάει για τεχνικά πρότυπα, technical standards στα αγγλικά, χωρίς όμως να λάβει υπόψη αυτά τα οποία προβλέπει η συνθήκη της Λισαβόνας. Βάσει της συμφωνίας με τους εισηγητές, σχεδόν εισηγητές για τα, την οδηγία Omnibus, εμείς έχουμε χωρίσει αυτές, αυτά τα πρότυπα σε δύο στοιχεία. Οι κανόνες για την μελλοντική κανονιστική εξέλιξη και αυτά που έχουν να κάνουν με την εφαρμογή. Αυτά βασίζονται στο 90 και, στο άλλα, και τα δεύτερα στο άρθρο 191 της συνδικής. Με την ε, συνδίκη της Λισαβόνας έχουμε μεγαλύτερες ευθύνες και αρμοδιότητες από ό,τι μας έδιναν προηγουμένως οι συνθήκες. Στην πρώτη περίπτωση μπορεί να τροποποιηθούν μονάχα από την Κομισιόν εάν υπάρξουν, εάν υπάρξει παραγνώριση βασικών κανόνων και για να αντιμετωπίσουμε αυτή τη μεγαλύτερη ισχύ που είχε η Κομισιόν για τα θέματα μεταρρύθμισης. Έχουμε δώσει στο Κοινοβούλιο περισσότερες ε, ε αρμοδιότητες, διότι βάσει των ρυθμίσεων για τις ε, κατεξουσιοδότηση πράξη θα πρέπει το Κοινοβούλιο να εμπλέκεται σε όλες τις περιπτώσεις που υπάρχει μια αλλαγή. Έχει φυσικά το δικαίωμα της αντίρρησης σε περίπτωση ε, κατεξουσιοδότηση πράξεων και μπορεί να αναστείλει τις εξουσίες κατεξουσιοδότηση στην Κομισιόν αν θεωρήσει ότι δεν τι χρησιμοποιεί σωστά η Κομισιόν. Επίσης περιλαμβάνουμε τροπολογίε που ζητούν μεγαλύτερη παρουσία σε αυτού που βρίσκονται στην ε, ομάδα ε, των τραπεζικών φορέων και σε ό,τι αφορά τι γενικέ κατευθύνσει, το ερώτημα είναι πώς θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ότι κάποιες αποφάσεις οι οποίες καταρχήν δεν έχουν κανονιστικό πλαίσιο αφορούν συστάσει και κατευθύνσει να έχουν το πιο δεσμευτικό δυνατό χαρακτήρα. Η φόρμουλα η οποία περιλαμβάνεται και σε πολλέ τροπολογίε και στο ενοποιημένο κείμενο βασίζεται σε τρει πυλώνες. Πληροφορία προ το Κοινοβούλιο σε σχέση με τι γενικέ κατευθύνσει που έχουν εγκριθεί, η πληροφορία του ποια είναι τα κράτη-μέλη τα οποία δεν έχουν τηρήσει αυτές τις κατευθύνσει ή τα θεσμικά όργανα, η δημοσίευση αυτών των αθετήσεων και μια ανάλυση όλων των μέτρων που θα πρέπει να αναλυθούν σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. Επειδή έχω και άλλους εισηγητές κοντά μου, δεν μπορούμε να επηρεάσουμε την ε, ελευθερία του τύπου, δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει, παραδείγματος χάρη, μια έλλειψη επαρκών κεφαλαίων σε, μια, σε ένα φορέα, γιατί αυτό θα δημιουργούσε προβλήματα. Επίσης ζητήσαμε να επανέλθει ο δεσμευτικός χαρακτήρας στην πρόταση τη Κομισιόν που δεν περιλαμβάνεται στο Συμβούλιο, ότι οι αποφάσεις του, του σώματος των ε, ρυθμιστών να εφαρμόζονται και όλα αυτά να κωδικοποιηθούν σε ένα κανονιστικό κείμενο το οποίο θα εφαρμόζεται πέραν των κανόνων εξέλιξης και των κανόνων εφαρμογής από τα όργανα τα οποία έχουν διασυνοριακές ε, λειτουργίες και συναλλαγές. Ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή είναι η εποπτεία των λεγόμενων συστημικών χρηματοπιστωτικών φορέων που λέγαμε στην αρχή φορείς ευρωπαϊκής διάστασης. Κατά αναλογία λοιπόν με φορείς οι οποίοι έχουν, έχουν ευρωπαϊκή σημασία και αυτούς που δεν έχουν άλλη σημασία. Έχουμε τονίσει δύο πράγματα στι εκθέσει. Καταρχήν ότι οι τωρινοί μηχανισμοί δεν μπορούν να λειτουργήσουν επαρκώ και πρέπει να του αλλάξουμε. Και δεύτερον, αυτή η αλλαγή είναι μονάχα δυνατή με το να εξυψώσουμε το εθνικό προφίλ τη εποπτεία ή να δώσουμε στην αρμόδια χώρα τη δυνατότητα να απαγορεύσει την χρήση θηγατρικών υποκαταστημάτων και θηγατρικών και δίνοντας ε, εξουσίες σε σχέση με τον έλεγχο της φερεγγιότητας των φορέων αυτών. Για παράδειγμα, χάρη, αυτό το οποίο κάνουν οι εθνικές ε, τράπεζες. Αυτή η απόφαση λοιπόν θα ήταν <clears throat> είναι αντίθετη με την ε, αρχή της ε, επικορικότητας. Έχουν γίνει πολλά πράγματα με την έκθεση. Πρώτα απ' όλα έχει λάβει χώρα η συνεδρίαση των G20 στο Πίτσπουργκ που ζήτησε μια ενδιάμεση συμφωνία για το πώ να εξασφαλίσουμε μια συμμετοχή του τραπεζικού τομέα στην επίλυση των προβλημάτων Αυτό Αυτή η έκθεση εμφανίστηκε πριν από λίγε μέρε και <clears throat> αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 4α όπου τονίζεται σαφώ ότι πρέπει να υπάρξει μια χρηματική συνεισφορά από τον τραπεζικό τομέα για να αντιμετωπιστούν οι περιοχέ κρίση. Στην Ευρώπη εμεί είχαμε μετά από την ε, έκθεση για τη στρατηγική 2020, η οποία ακολουθεί την ίδια φιλοσοφία, ότι ζητούμε από τον τομέα αυτό να επομιστεί το κόστος της κρίσης, ώστε να μην πρέπει να πληρώσουν οι φορολογούμενοι. Και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 25ης-26ης Μαρτίου μίλησε για τα συστημικά ιδρύματα ως μια σημαντική κατηγορία για να μπορέσει να υπάρξει ένα καθεστώς στον τραπεζικό τομέα έχετε διαβάσει φαντάζομαι τον οικονομικό τύπο όπου υπάρχει η ίδια αυτή η συζήτηση που γίνεται εξάλλου και στο, στο Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών όπου επειδή δεν συμφώνησαν οι Ρεπουμπλικάν και ακολούθησαν μια παρελκυστική τακτική δεν, εξε, ε, ενεκρίθη αυτή η ρύθμιση. Πώς θα προχωρήσουμε τώρα καταρχήν σε σχέση με την αρχική έκθεση, με τις αρχικές εκθέσεις των τεσσάρων ε, <clears throat> εισηγητών εφαρμόσαμε την λογική ότι πρέπει να έχουμε ευρωπαϊκή εποπτεία για ευρωπαϊκού φορεί. Για να είναι αποτελεσματικό το σύστημα, να μην έχουμε περισσότερη γραφειοκρατία και να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε το δυνατόν την γνώση που είχαν οι εθνικοί ρυθμιστέ, έχουμε πει με απόλυτη σαφήνεια ότι η Ευρωπαϊκή Αρχή θα μπορέσει να εξασκήσει αυτή την εποπτεία μόνο μέσω των εθνικών εποπτών με μία σχέση η οποία θα εξασφαλίσει ότι θα ακολουθούν τις δομές της Ευρωπαϊκής Εποπτείας και θα υπάρχει κατακαιρματισμός των προτύπων και ετερογένεια του τρόπου εποπτείας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Για να καθορίσουμε ποιοι είναι οι συστημικοί φορείς, χθε. <clears throat> και αυτό βρίσκεται στο ενημερωμένο κείμενο, δεν ξέρω ποια μορφή θα λάβει. Υπάρχει μια πρόταση των φιλελευθέρων της Σιλβί Γκουλάρ, η οποία περιλαμβάνει και το προφίλ του κινδύνου μέσα στην κατηγοριοποίηση των πιστοτικών ιδρυμάτων. Γιατί δεν είναι μονάχα θέμα μεγέθους για να δούμε το θέμα του κινδύνου, αλλά το επιχειρηματικό μοντέλο, η έκθεση σε κινδύνους και η αλληλοσύνδεση διαφόρων πιστοτικών ιδρυμάτων. Υπάρχει στη ρήτρα αναθεώρησης η διατύπωση ότι έξι μήνες μετά από την θέση εφαρμογή αυτού του κανονισμού θα πρέπει να μας δώσει τις προτάσεις κανονισμού, τις κανονιστικές προτάσεις οι οποίες θα συμπληρώσουν το πλαίσιο το οποίο διαγράφεται με τις τωρινέ <clears throat> αποφάσεις. Επίσης αναφέρεται ότι πρέπει να υπάρχει ένας φορέας για την επίλυση των διαφορών, κάτι το οποίο έρχεται αμέσως από την έκθεση Ελίζα Φερέιρα. Πρόκειται στο να έχουμε ένα φορέα μέσα στο, θεσμικό φορέα, ο οποίο μπορεί να παρακολουθήσει μια κρίση από τη στιγμή που ξεκινάει μέχρι τη στιγμή που τελειώνει και θα μπορέσει να αναλάβει όλε τι αποφάσει που θεωρεί σκόπιμε για την ε, παροχή εγγυήσεων, για τη δανειοδότηση κτλ. Και επίση προβλέπεται με συμφωνία όλων των συζητητών και με την σύμφωνη απόψη των περισσότερων τροπολογιών ότι θα πρέπει να αποφύγουμε με κάθε τίμημα το λεγόμενο ηθικό κίνδυνο. Η διάσωση λοιπόν θα πρέπει να γίνει μονάχα εάν δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα. Καθορίζεται λοιπόν εξασφάλιση των καταθέσεων που έχει να κάνει με την ε, μορφή των θεσμικών ιδρυμάτων. Δεν ε, μπορούμε να δεχτούμε την πρόταση να υπάρχει διαφορετική κάλυψη σε εθνικό επίπεδο όταν κυκλοφορούν ελεύθερα τα κεφάλαια και επίσης δημιουργείται και ένα ταμείο διάσωσης το οποίο προχρηματοδοτείται από τις εθνικές αρχές και αυτό ε, διαμορφώνεται με βάση το επίπεδο κινδύνου και τη βάση μιας σειράς κριτηρίων, το λεγόμενο dashboard, το, η επιφάνεια ελέγχου για να δούμε πώς θα πρέπει να αντιμετωπιστούν αυτά τα θέματα. Υπάρχει επίσης το, το κείμενο το οποίο αφορά τις ασφάλειες των ασφαλιών, το οποίο το υποστήριξε και η κυρία Λούλινγκ εδώ. Ο κανόνας εδώ είναι ότι θα λαμβάνει αποφάσεις με απλή πλειοψηφία και μόνο για τις αποφάσεις που έχουν κανονιστικό χαρακτήρα θα χρησιμοποιείται η ειδική πλειοψηφία, γενικέ κατευθύνσει, αυτέ επίση οι οποίε έχουν αντίκτυπο στον προπολογισμό. Σε ό,τι αφορά την ρήτρα τελική ευθύνη, έχουν γίνει πολλέ τροποποιήσει σε σχέση με το αρχικό κείμενο. Η μεγάλη πλειοψηφία των βουλευτών παρουσίασαν τροπολογίε όπου δεν δείχνουν μεγάλη υποστήριξη στο ότι ένα κράτο μέλο θα μπορούσε να λάβει μια απόφαση η οποία αφορά ένα συγκεκριμένο ρυθμιστή. Και εάν δεν υπάρξει μια συμφωνία να φέρουν το θέμα αυτό στο Συμβούλιο με δυνατότητα αναστόλης από την πλευρά του, του Συμβουλίου. Αυτό είναι μια λαθασμένη διαδικασία. Αν υπάρξει ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα το οποίο ε, πτωχεύει, αυτό θα μολύνει και τα υπόλοιπα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Θεωρούμε ότι ένα κράτο μέλο το οποίο λέει ότι μια απόφαση έχει αποτέλεσμα στον προπολογισμό θα πρέπει να το επιχειρηματολογήσει, να το βασίσει, να το δείξει με μια οικονομική μελέτη η οποία εκτιμά και αποτιμά αυτόν τον κίνδυνο για τον προπολογισμό και να υπάρχει το τεκμήριο νομιμότητος των αποφάσεων που λαμβάνονται από τους εθνικούς ρυθμιστές και απαιτείται μια ειδική πλειοψηφία για να διατηρηθεί η απόφαση η οποία έχει ληφθεί, για να ανατραπεί αυτή η απόφαση θα είναι απαραίτητο να υπάρξει μια ειδική πλειοψηφία, μια ενισχυμένη πλειοψηφία. Και στις ε, δύο περιπτώσεις το κράτος μέλος το οποίο έχει ζητήσει την εφαρμογή αυτής της ρήτρας δεν θα συμμετέχει στις ψηφοφορίες. Μια τελική αίτηση, όπως είπα και προηγουμένως, σας έχω δώσει το κείμενο με την ενοποιημένη μορφή της κάνοντας τις ε, απαραίτητες συμβιβαστικές τροπολογίες όπου αυτό ήταν απαραίτητο. Φυσικά το κείμενο αυτό έχει ένα προσωρινό χαρακτήρα, θα ξεκινήσουμε τη διαπραγμάτευση και θα συνεχιστεί και σήμερα και αργότερα η διαπραγμάτευση μεταξύ των ε, ε, εισηγητών, μέχρι ότου η πρόεδρος θεωρήσει ότι είναι όριμα τα πράγματα να καταλήξουμε σε μια ψηφοφορία μεταξύ της ψηφοφορία στην Επιτροπή μα και τι Ολομέλειε, μπορούμε ίσω να χρησιμοποιήσουμε τον χρόνο για να κάνουμε περαιτέρω διαπραγματεύσει και η μεγαλύτερη διαπραγμάτευση θα γίνει όταν το Κοινοβούλιο έχει ήδη λάβει την απόφασή του και θα πρέπει να διαπραγματευτούμε με το Συμβούλιο. Γι' αυτό σα ζητώ σε εκείνε τι στιγμέ να μπορέσουμε να κρατήσουμε μια στεναρή και ισχυρή θέση ενώπιον του Συμβουλίου, μια ενωμένη στάση, γιατί αυτέ οι διαπραγματεύσει, όπω είναι πάντα παράδοση, εγώ θα επανέλθω και θα συζητήσω μαζί σας για να κλείσουμε όλα τα απαραίτητα συμπεράσματα. Αλλά σας ζητώ να προχωρήσουμε με τον ταχύτερο δυνατό τρόπο ώστε να προχωρήσουμε και να εκ... θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου και προς την γραμματεία για το τιτάνιο έργο στο οποίο έφερε σε πέρας. Ποιες είναι τώρα οι τροπολογίες που θεωρούμε ότι μπορούν να αποσυρθούν και ποιες είναι αυτές οι οποίες θα πρέπει να διατηρηθούν μπορούμε να παραμείνουμε σε επαφή για να δούμε αν αυτές οι τροπολογίες διασπούν την φιλοσοφία που διατρέχει τις εκθέσεις, κάτι το οποίο χρειάστηκε πολύ χρόνο για να το εδραιώσουμε. Έχουμε αντιμετωπίσει θέματα τα οποία στο παρελθόν δεν τα είχε σκεφτεί κανένα και τώρα πράγματι τα αντιμετωπίσουν όλα. Ο Επίτροπο Παρνιέ στο Συμβουλιακό ΦΥΝ έχει προτείνει το θέμα αυτό του Ταμείου Διάσωση. Εμεί το είχαμε αναφέρει ήδη στο παρελθόν. Υπάρχουν λοιπόν πολλά σημεία στα οποία συμφωνούμε με την Επιτροπή, υπάρχουν άλλα θέματα τα οποία είναι εκκρέμη και ελπίζω ότι θα μπορέσουν να διαλευκαθούν όλα αυτά σε ένα έφθετο χρόνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε και θέλω να ευχαριστήσω όλου αυτού οι οποίοι καταστάν τροπολογίε για την προσπάθεια την οποία κατάβαλαν για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε μια έκθεση, ένα θέμα το οποίο ήταν πάρα πολύ μεγάλη σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδίω στι δύσκολε στιγμέ, οποίε διατρέχουμε πάρα, πάρα πολύ. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα ακολουθήσουμε τη σειρά των εισηγητών τώρα στι αγορεύσει. Ε, ο Σβέν για την αρχή για τις αγορές. Μπορώ, δεν μπορώ να παρά να επαναλάβω εν συντομία αυτά που είδε, ήδη είπε ο συνάδελφος Ζε Μαρία Μαργάιο ότι υπάρχει πολύ καλή συνεργασία μεταξύ των διαφόρων εισηγητών με τη γραμματεία, με τους διάφορους σκιώδεις πρέπει να πω ότι μεθοδολογικός πώς ε, αυτό αποτελεί πρόκληση. Έχουμε τρεις εκθέσεις που είναι πολύ κοντά η μία στην άλλη. Δεν, δεν μπορεί να διαφέρουν σημαντικά, αλλιώς θα ήταν γελίο, δεν θα υπήρχε συνοχή. Ταυτόχρονα οι τρεις εκθέσεις πρέπει να συνδεθούν με τη δουλειά για το ESRB, άρα χρειάζεται συνεκτικό πλαίσιο. Και αν συναντηθούν οι συγητέ και οι σκιώδει σε μια συνεδρίαση, ποτέ δεν καθορίζεται μια προθεσμία και η συνεδρίαση πιθανότατα δεν θα οδηγήσει πουθενά. Είναι πολύ δύσκολο να μιλήσει κανείς με όλους που συμμετέχουν. Για μένα, σαν εισηγητή για το ΕΣΜΑ, πρέπει να συζητήσω με αυτούς που είναι υπεύθυνοι για το ΕΜΠΑΡ, για το ΑΙΟΠΑ και λοιπά, με του άλλου γιατί είναι αλληλένδετα όλα τα θέματα. Είναι αδύνατο να συζητήσω με όλου σε λεπτομέρειες, άρα είναι θέμα ποιότητα πληροφοριών, ποιότητας ανταλλασσομένων πληροφοριών μεταξύ συγχυτών. Στη συζήτηση λοιπόν θα ήθελα το εξή. Θέλουμε να αλλάξουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι προφανές αυτό, διότι πευλήθησαν τροπολογίες αν διαφωνεί όμως κανείς με τροπολογίες που υπευλήθησαν από άλλους ή από τους εισηγητές, δεν είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Και η όλη διαδικασία μπορεί να γίνει χαόδης. Στη συζήτηση παρακαλώ να δηλώσετε σαφώς που διαβλέπετε δυσκολίες, προβλήματα στη διαδικασία. Και επιθεματων επί των οποίων δεν μπορέσετε να υποβάλλετε τροπολογίες, που όμως ίσως οδηγήσουν σε απρόβλεπτα αποτελέσματα όσον αφορά τις ε, ψηφοφορίες. Και δεν υπάρχει δυνατότητα να συζητήσουμε με τον προτέρων όλες λεπτομέρειες. Γι' αυτό ας ανοιχτοί συνάδελφοι. Για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα και των προτέρων. Είμαι ανοιχτό για άμεσε ανταλλαγέ απόψεων με οποιοδήποτε από εσά, έστω και αν δεν είστε σκιώδη εισηγητή. Για τι τροπολογίε. Θα αναφερθώ στους βασικότερους τομείς που υπευλήθησαν όσον αφορά την Ευρωπαϊκή αυτή του για τίτλους ΕΣΜΑ. Υπάρχει γενική συνένεση για την προστασία των επενδυτών, ισότιμες συνθήκες για όλους, δυνατότητα διαιτησία όσον αφορά τον έλεγχο και οικονομική ανάλυση του τομέα που πρέπει να είναι στόχος του φορέα της ΕΣΜΑ. Υπευλήθησαν και κάποιες τροπολογίες για την σύνθεση της ομάδας των ενδιαφερομένων μερών. Δεν υπάρχουν διαφορές εδώ. Η συζήτηση για τη ρήτρα διαφύλαξης αναφέρθηκε ήδη. Δεν επαναλαμβάνω τα υποθέτα. Για το άρθρο 7, τεχνικά πρότυπα, υπήρξαν πολλές τροπολογίες. Δεν υπάρχουν μεγάλες διαφορές. Για τις άμεσες εξουσίες, άρθρο 8 ως 11, υπήρχαν κάποιες διαφορές, αλλά η πλειοψηφία επιθυμεί μεγαλύτερη αύξηση των εξουσιών αυτών. Για κατεπίγους ανάγκη, ποιος διακηρύσει ότι έχουμε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Εγώ είμαι υπέρ του ότι η ESRB θα πρέπει να δηλώνει ότι έχουμε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Αλλά οι εξουσίες πρέπει να ανακοινώνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για νομικούς λόγους. Πρέπει να επιλεχθεί αυτή η λύση. Για την άμεση εποπτεία. Υπάρχουν διαφορετικές θέσεις. Συζητήθηκαν όλα, δεν τα επαναλαμβάνω για την άμεση εποπτεία στην έκθεσή μου για τους οίκους συμψηφισμού υπάρχουν διαφορές. Είμαι υπέρ της άμεσης εποπτείας από πλευράς ΕΣΜΑ, της αρχής για, τους, ε, τις αγορές τίτλων. Θα πρέπει να υπάρχει και δυνατότητα απαγόρευσης κάποιων συναλλαγών. Στην κατάσταση που είμαστε τώρα, Βλέπουμε ότι η ΕΣΜΑ θα πρέπει να έχει αυτές τις εξουσίες. Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται αυτές οι εξουσίες συχνά, θα πρέπει να είναι μια δυνατότητα σε κάποιες περιστάσεις. Τέλος, το θέμα του ε, Συμβουλίου Εφέσεων, του Φορέα Εφέσεων, προσωπικά, δεν ξέρω κατά πόσο αυτός ο φορέας είναι νόμιμος και αν είναι καλός τρόπος καλή λύση. Κατά πόσο είναι νόμιμη προσέγγιση να αμφισβητηθούν οι λιμένες αποφάσεις. Και αν δικαιολογείται δημοκρατικά αυτή η προσέγγιση. Ευχαριστώ όλους εκ νέου και με τα χαράς να ακούσω τα σχόλιά σας. Ευχαριστώ. Λείπει ο Πέτρος Σκίνερ και θα αντικατασταθεί Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πράγματι, εγώ θα τον αντικαταστήσω. Θέλω να κάνω δύο σχόλια. Πρώτον, θα σκιαγραφίσω τη θέση του εισηγητού και δεύτερον, αν μου το επιτρέπετε, θα ήθελα να κάνω και δικά μου σχόλια ως συντονιστής για τους σοσιαλιστάς και δημοκράτας. και ως προς το μέλλον. Λοιπόν, ο Πέτρος Σκίνερ είναι υπεύθυνο για τον τομέα των ασφαλίσεων. Έχει όμως ανηλυμένες υποχρεώσεις και δυστυχώς λείπει σήμερα. Δυστυχώς. Mm. Στα άρθρα με ένα μέχρι 20 ζητάει ο Σκίνερ να υπάρξει ένας νέος ορισμός και να επεκταθεί το ευρωπαϊκό σύστημα εποπτείας περαιτέρω. Είναι επίσης υπέρ της ενίσχυσης του ρόλου nationalen Autoritäten zu unterstützen, wo es darum geht, das Stresstesting και θα θέλαμε να καταλήξουμε σε μια κοινή μεθοδολογία και για την ΕΣΜΑ και για την ΣΕΣΡΜ. Υπάρχει, τίθεται και ένα θέμα νομιμότητας εδώ και κατά πόσον μπορεί και πρέπει να γίνει εποπτεία ανατομέα. Προτεραιότητα δίνει σε αυτό ο κύριος Σκίνερ. Αυτό όμως στο οποίο αντιτίθεται και επιμένει σε αυτό είναι να αποδυναμωθεί η ΕΣΜΑ. Όπως διαφαίνεται από το σύστημα, η ΕΟΠΑ μάλλον, από το Συμβούλιο, όπως διαφαίνεται από τις τελευταία συμπεράσματα του Συμβουλίου. δείχνει επίσης μεγάλη φρόνηση ως προς τη διατύπωση που πρέπει να έχει το κείμενο. Όταν λοιπόν οι εκτιμήσεις αυτές δεν είναι επαρκείς, αναφέρεται το στα αγγλικά unnecessary markup of language, δηλαδή ότι υπάρχει μια περιττή χρήση διατυπώσεων η οποία δεν βοηθάει ιδιαίτερα. Το άρθρο 22 υποστηρίζει την δημιουργία δύο ομάδων εμπλεκομένων, καταρχήν για, την, ε, για το σύστημα συντάξεων και το άλλο για τα θέματα ασφαλίσεως, ασφαλιστικές εταιρείες. Εγώ θεωρώ ότι είναι μια καλή ισορροπία εδώ, μεταξύ των δύο αυτών ομάδων εμπλεκομένων και πιστεύω ότι είναι απαραίτητο να διατηρήσουμε και τη δυνατότητα αυτές οι ομάδες να εκφράζουν την άποψή του ακόμα και σαν μειοψηφίε. Αυτό το οποίο εγώ δεν υποστηρίζω είναι η πλευρά του, ε, του οικονομικού κλάδου, οι εταιρείε δηλαδή, να εκπροσωπούνται υπερμέτρως. Το άρθρο 23, η ρήτρα διαφύλαξης, ζητά εδώ να υπάρχει από τα κράτη-μέλη μια έκθεση αντικτύπου και να μπορούν με τον τρόπο αυτό να ε, εφαρμόσουν τις αποφάσεις της ΑΙΟΠΑ, του φορέα αυτού λοιπόν για τις ε, ασφάλειες και τις ε, συντάξεις. Αυτό είναι χρήσιμο λοιπόν να αντιμετωπιστεί και να μην οδηγήσει σε περαιτέρω προσκόμματα σε ό,τι αφορά την πολιτική. Τα άρθρα 25 έως 38 τώρα επίσης για την ΑΙΟΠΑ, για τον φορέα για τις συντάξεις και τις ασφάλειες, υποστηρίζει ότι ο ρόλος του, μάλλον, ο πρόεδρος θα πρέπει να καθορίζεται από ένα, τομή, από ένα συμβούλιο εποπτικό και υποστηρίζει το ότι θα πρέπει να υπάρχουν κατά πλειοψηφία λήψεις αποφάσεων σε όλες τις σημαντικές αποφάσεις στο, ταμείο, στο Συμβούλιο των Εποπτών Αυτό το οποίο όμως δεν υποστηρίζω είναι να δημιουργηθεί ένα ανεξάρτητο πάνελ από εμπειρογνώμονες, γιατί αυτό θα δημιουργήσει περαιτέρω γραφειοκρατία. Για, τις, για τα άρθρα 39 43 που αφορούν το Εποπτικό Συμβούλιο, αυτό έχει να κάνει με το να τεθεί όλη αυτή η εποπτική αρχή στην Φραγκφούρτη. Τα άλλα θέμα, το άρθρο 44 και επέκεινα, υποστηρίζουν το να υπάρξει μια περαιτέρω διευκρίνηση και αξιόπιση του ρόλου της ε, ΣΑΙΟΠΣ και η δημιουργία της ε, Εποπτικής Αρχής για την Ασφάλεια και τις Επαγγελματικές Συντάξεις και τονίζω ότι είναι απαραίτητο και χρήσιμο να υπάρχει και συμμετοχή εκπροσώπων από τρίτες χώρες. Συνοπτικά και καταληκτικά, ο εισηγητής πιστεύει ότι θα πρέπει να υπάρχει μια ισχυρή δομή στην ε, ΑΙΟΠΑ, στην ε, Αρχή για τις Επαγγελματικές Συντάξεις και την Ασφάλεια, ώστε να μπορέσουμε με τον τρόπο αυτό να εξασφαλίσουμε ιδιαίτερα τα ζητήματα άμεση εποπτείας για το κατά πόσον πρέπει ορισμένα προϊόντα να απαγορευτούν και επίσης στο να υπάρχει μια διαδικασία λήψης απόφασης για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε εδώ την εφαρμογή ορισμένων προτάσεων της κυρίας Φερέρα και άλλες προτάσεις οι οποίες ενδεχομένως να προκύψουν από την Κομισιόν. Πιστεύω εν ότι η θέση αυτή όπως ε, παρουσιάζεται από το έγγραφο είναι μια θέση Ο συντονιστής λοιπόν της ομάδας μου θέλησα να παρουσιάσω τη θέση της ομάδας μου. Νομίζω ότι η Επιτροπή μας έχει αναλάβει ένα ιδιαίτερα φιλόδοξο εγχείρημα. Ο στόχος μας είναι να δώσουμε στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μια απάντηση στην πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση με οποία προκάλεσε η χρηματοοικονομική κρίση. Κυρία Πρόεδρε, εγώ θέλω να τονίσω ότι κατά την άποψή μου όλοι οι εμπλεκόμενοι, οι εισηγητές και σκιώδες οι εισηγητές έχουν κάνει ένα ιδιαίτερα υπεύθυνο και υψηλού επίπεδου έργο. Δεν είναι εύκολο να καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα, γιατί έχουμε διαφορετικές απόψεις τόσο σε ό,τι αφορά και μέσα στις δικές μας πολιτικές ομάδες, αλλά και μεταξύ των πολιτικών ομάδων. Και φυσικά δεν μπορεί να είναι διαφορετικό, διότι οι θέσεις οι οποίες εκπροσωπούνται από εμά είναι όλες έγκυρες. Δεν θέλω να σχολιάσω αυτά τα οποία λέει ο κύριος Σκίνερ. Πιστεύω ότι όλες οι προσπάθειές μας βασίζονται στην δική μας εμπειρία που είχαμε στις χώρες μας με τον χρηματοπιστωτικό τομέα, που είναι διαφορετικές φυσικά αυτές οι εμπειρίες. Πιστεύω λοιπόν ότι όλες αυτές οι προσπάθειες έχουν σημαντική αξία και είναι τώρα απαραίτητο με γαλήνη και με συγκέντρωση να μπορέσουμε να συνεχίσουμε αυτό το εγχείρημα προς όφελος των φορολογουμένων. Θέλω να πω κάτι ακόμα όμως γιατί βρισκόμαστε στην τελική φάση της προετοιμασίας του έργου αυτού. Εγώ υποστηρίζω ιδιαίτερα να εστιάσουμε ακόμα περισσότερο την προσοχή μας στα θέματα αυτά, ώστε να μπορέσουμε να επιτύχουμε μια μεγαλύτερη σύγκληση απόψεων, ώστε να έχουμε μια όσο δυνατόν μεγαλύτερη συνένεση στην Επιτροπή μας και ότι στο βαθμό του δυνατού να σταθούμε στις διάφορες ιδιαιτερότητες οι οποίες μπορεί να υπάρχουν μεταξύ διαφορετικών κλάδων. Ο κύριος Σκίνερα, παραδείγματος χάρη, λέει ότι ορισμένα πράγματα σε ό,τι αφορά τον τομέα των ασφαλιστικών εταιριών, από τι ασφαλιστικέ εταιρείε, υπάρχει μια διαφορετική οπτική γωνία από ό,τι από την πλευρά των τραπεζών. Πιστεύω όμω ότι σε αυτή την τελική ε, φάση δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό από το να, να υπάρξει και σύνδεση με τις πολιτικές απόψεις των κομμάτων μας, γιατί είναι απαραίτητο η τόσο δύσκολα και με τόση προσπάθεια επιτευχθεί σε συμφωνίες να εγκυροποιηθούν και να γίνουν δεκτές και από τους συναδέλφους μας στα πολιτικά κόμματα. Γιατί τελικά δεν είναι μονάχα θέμα επιτυχούς εργασίας αλλά και σωστής επικοινωνίας με τους συναδέλφους μας. Και θα ήθελα λοιπόν να συζητήσουμε αυτό το θέμα και στους συντονιστές ότι αν προκύψει μια κατάσταση που θα πρέπει να επιλέξουμε μεταξύ του να έχουμε ένα καλό προϊόν ή να έχουμε ταχύτητα στη διεκπαιρέωση. Εγώ προτιμώ να έχουμε ένα καλό προϊόν, ακόμα και αν αυτό καθυστερήσουμε, αν χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο. Αν γίνει σαφέ ότι χρειάζεται περισσότερο χρόνο λοιπόν, για την εκπόνηση αυτών των εκθέσεων και να καθυστερήσουμε τη διαδικασία τη απόφαση, εγώ συμφωνώ, γιατί για μένα, για τη δική μου άποψη, είναι το σημαντικότερο το να έχουμε ένα καλό τελικό αποτέλεσμα και είναι δευτερεύον να δράσουμε ταχαίω. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. Um, now we'll... Ευχαριστώ πολύ. Η Σιλβί Γκουλάρ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εντάχει. Διότι εργαζόμαστε συλλογικά, δεν θα επαναλάβω αυτά που υπόθηκαν. Έχουμε υψηλό επίπεδο φιλοδοξιών. Θα προσπαθήσουμε να εργαστούμε το ταχύτερο δυνατόν, χωρί να επηρεάσουμε όμω αρνητικά την ποιότητα τη ουσία. Θα ήθελα να προβώ σε τρία σχόλια όσον αφορά το κείμενό μου. Ευχαριστώ καταρχά εκείνου που έβαλαν επικοδομητικέ τροπολογίε. Κάναμε συνεδρίε των σκιωδών πρόσφατα. Η γραμματεία, την οποία ευχαριστώ, έκανε πάρα πολύ δουλειά. Πιστεύω ότι δεν είμαστε μακριά από κάποια συμφωνία. Τα δύο εκρεμή σημεία είναι ο βαθμός εν γέννη ελέγχου από τις κεντρικές τράπεζες, ποιος είναι ο βαθμός ανοίγματος, υπάρχουν τροπολογίες υπέρ της κεντρικής τράπεζας και τροπολογίες υπέρ του μεγάλου ανοίγματος που να δούμε τη μέση λύση και ο βαθμός της διαφάνειας μετά είναι ευκταίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Συστημικού Κινδύνου να δημοσιοποιεί τις αποφάσεις της, είναι πιο αποτελεσματικό να μπορεί να απειλεί να δημοσιεύει. Δεν θα επιστρέψω σε λεπτομέρειες. Θέλω να ακούσω ε, εσάς που έχετε κάποια σχόλια. Ο συσχετισμός με τις άλλες ε, εκθέσεις πρέπει να ομολογήσω ότι υπάρχει ε, ότι θέλω να πω ότι εκτελήσω διεργασίες. Όπως είπε ο Χωσέ Μανουέλ, δεν έχουμε ολοκληρώσει εργασίες. Υπάρχει ένα βασικό θέμα Δηλαδή, βάσει ποιων κριτηρίων οι αρχές παρεμβαίνουν άμεσα ε, επί κάποιων ε, ιδρυμάτων. Είναι το πιο περίπλοκο θέμα. Δεν είναι πολιτικό θέμα. Είναι ένα θέμα του να καθορίσουν σε ποιο βαθμό είναι ένα δίκτυο εθνικών αρχών και κανείς δεν θέλει να τα θέσει όλα σε κεντρικό επίπεδο και σε ποιο βαθμό όμως από καιρούς καιρών θα μπορούμε να παρεμβαίνουμε στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Να πω αυτά που είδα στην κυρία Φερέρα για την έκθεσή της και λοιπά, ότι έχω κάποια αμφιβολία κυρίως όταν σκέφτομαι τις ακροάσεις που οργανώσαμε. Όσον αφορά το εξής, δηλαδή να καθορίσουμε κάποια ιδρύματα, κάποιους θεσμούς ε, που έχουν συστημικό χαρακτήρα. Η κρίση απεδείξε ότι τα ιδρύματα ενός μεγέθους μετρίου μπορούν να παρουσιάζουν κάποιο κίνδυνο. Μετά, σύμφωνα με όλου του ειδικού που ακούσαμε και του τομέα των ασφαλίσεων και των τραπεζών και της αγοράς, ο συνδυασμός κάποιων κριτηρίων είναι που δημιουργεί τον κίνδυνο και όχι απλώς το μέγεθος του Ιδρύματος. Και τρίτον, εγώ είμαι πολύ ευαίσθητη όσον αφορά τα θέματα του θεμητού ανταγωνισμού. Εάν έχουμε έναν κατάλογο ε, εγκατεστημένων συστημικών Ιδρυμάτων που παρουσιάζουν κίνδυνο, μπορεί να ξεχάσουμε κάποιους φορείς και να δημιουργήσουμε στρεβλώσεις ανταγωνισμού, τεράστιες στρεβλώσεις Οπότε σταματώ εδώ, είναι βασικό θέμα της εκθέσεως και της εκθέσεως της κυρίας Φερέρα και ένα σημείο κλειδί όλων των προσπαθειών που κάνουμε για τη βελτίωση εποπτείας. Εγώ δεν ισχυρίζομαι ότι ε, ξέρω ποια είναι αλήθεια. Κάναμε ακροάσεις, συζητήσαμε με διάφορους πανεπιστημιακούς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει διαφορετική άποψη. Υπάρχει και μία μόδα, λοιπόν. Ε, αυτή των θεσμών των συστημικών. Είναι κάτι που βγήκε από τα συμπεράσματα του Συμβουλίου. Και η μόδα είναι αυτά τα... η ανοιξιάτικη μόδα είναι αυτά τα συστημικά ιδρύματα. Θα πρέπει να προσέξουμε να μην βρούμε μια λύση η οποία τελικά να κινδυνεύσει να αποβεί αντιπαραγωγική. Αυτά και ευχαριστώ. Ευχαριστώ λέει Πρόεδρος. Ρεμό, θες να πεις κάτι? Όσον αφορά τη λειτουργία, είναι πολύ σύντομη η εκθεσή μου, οπότε 30 δευτερόλεπτα χρειάζομαι. Να πω ότι έλαβα μόλις 12 τροπολογίες. Είναι πολύ εύκολο να ληφθούν οι υπόψεις στο κείμενο, δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα, ευχαριστώ. Οπότε χρησιμοποιήστε το χρόνο τώρα για τη συζήτηση με θέμα της μεγάλες εκθέσεις. Ευχαριστώ πολύ. Για το Omnibus 1 Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Η Γενικού Περιεχομένου 1, η Omnibus 1 λοιπόν, έχει, παρου, έχει δεχτεί μια σειρά από τροπολογίε, ο οποίο θέλω να ευχαριστήσω όλου αυτού που κατέθεσαν τροπολογίε. Δεν είχα την προηγούμενη ευκαιρία της, την ευκαιρία να συναντηθώ μαζί του για να ανταλλάξουμε απόψει, αλλά σήμερα το απόγευμα θα του στείλω την δική μου κρίση για τι τροπολογίε και τι προτάσει μου για συμβαστικέ τροπολογίε. Έχουμε λοιπόν αυτές τις 114 τροπολογίες. Καταρχήν, εγώ θα διατυπώσω 28 συμβασικές τροπολογίες, οι οποίες νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό συμπληρώνουν και συνοψίζουν αυτές τις ε, τροπολογίες. Εγώ υποστηρίζω σε μεγάλο βαθμό περίπου 50 από τις τροπολογίες οι οποίες έχουν κατατεθεί και είναι μονάχα 18 τροπολογίες, τις οποίες εγώ έχω σημαντικές αμφιβολίες, κυρίως γιατί δεν εξασφαλίζουν τη συνεκτικότητα με το σύνολο της έκθεσης, επομένω η συμπερίληψή του θα μπορούσε να αποδυναμώσει το σύνολο τη δομή που περιέχει η έκθεση αυτή. Οι περισσότερες τροπολογίες αφορούν τις οδηγίες για τις ε, αγορές ε, χρηματιστηριακού χαρακτήρα, για τη MIFID και για τα διαφημιστικά φυλάδια. Επίσης έχουν παρουσιαστεί πολλές τροπολογίες σε ό,τι αφορά τις κεφαλουχικές απαιτήσει. Η άποψη που εγώ ακολουθώ σε ό,τι αφορά την ε, αξιολόγηση των, τροπολογιών αυτών και τις προτάσεις που θα παρουσιάσω είναι καταρχήν πιστεύω ότι θα πρέπει να διατηρήσουμε μια συνοχή μεταξύ της οδηγίας όμνιμους και του συνόλου των κανονισμών που θεσπίζουν τις βασικές αρχές. Θα πρέπει να μεταφέρουμε τις νέες αυτές ε, συμφωνίες και κανονισμούς στις νέες οδηγίες. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε επομένω την συνεκτικότητα με το σύνολο του πακέτου εποπτείας και δεύτερον όλες αυτές οι πρότασεις οι οποίες έχουν σαν στόχο το να ενισχύσουμε το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη διαδικασία οικονομικής ανάπτυξης αυτών των οικονομικών οδηγιών, θα πρέπει να λάβουμε πάντα υπόψη μας ότι εμείς θα πρέπει να τις υποστηρίξουμε. Και επίσης είναι απαραίτητο να ενημερώσουμε και βάσει τη συνθήκη της Λισαβόνας εξουσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Υπάρχουν πράγματα τα οποία υπάρχουν σε δυνητικό επίπεδο. Είναι το να έχουμε πρότυπα σε νομικό επίπεδο και είναι διαφορετική κατάσταση με τις τεχνικές, ε, τα τεχνικά πρότυπα. Έχουμε τη διαδικασία κατεξουσιοδότηση πράξεων που εφαρμόζονται με τον έλεγχο του Κοινοβουλίου και η άλλη διαδικασία είναι αυτές που γίνονται με εκτελεστικές αποφάσεις. Εμείς θα πρέπει να κατατάξουμε λοιπόν αυτά τα οποία θέλουμε τα πρότυπα σε μία ή την άλλη κατηγορία. Πιστεύω ότι αυτά που έχουν να κάνουν με τις τεχνικές ρυθμίσεις να υπάρχει κάποια συμφωνία για να προχωρήσουν χωρίς να γίνεται αυτό στο περιθώριο των συνδικών και χωρίς έλεγχο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τρίτον, όλα αυτά που έχουν να κάνουν με έγκριση για μεταρρύθμιση, όλα αυτά που έχουν να κάνουν με ενημέρωση μάλλον οδηγιών οι οποίε θα πρέπει να αναθεωρηθούν. Αυτέ οι τροπολογίε είναι καλόδεκτε. Πιστεύω ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη όμω εδώ και τα χρονοδιαγράμματα. Σε ορισμένε περιπτώσει, οι τροπολογίες αυτέ ζητούσαν συγκεκριμένα χρονικά πλαίσια για να παρουσιάσει προτάσει μεταρρύθμιση τη Κομισιόν και για τα τεχνικά πρότυπα εγώ χαιρετίζω και υποδέχομαι θετικά όλε αυτέ τις τροπολογίε. Υπήρξαν επίση ορισμένες τροπολογίες που έχουν να κάνουν με ευαίσθητα θέματα όπως είναι το υβριδικό κεφάλαιο, είναι θέματα τα οποία πρέπει να αρχίσουμε να τα επεξεργαζόμαστε και έχουμε εδώ ένα πολύπλοκο κανονιστικό πλαίσιο το οποίο πρέπει να καταλήξουμε και εγώ συμφωνώ ότι θα πρέπει να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία αλλά συγχρόνως το όριο του 2014 που έχουμε θεσπίσει προηγουμένως θα πρέπει να διατηρηθεί για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε περισσότερο στην εφαρμογή κεντρικών προτύπων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τέλος, αυτό το οποίο θέλω να τονίσω είναι ότι όλες αυτές οι τροπολογίες είναι καλόδεκτες, νομίζω ότι είναι σημαντικές βελτιώσεις στο κείμενο και υπάρχει και μια άλλη αντιμετώπιση την οποία έχω <clears throat> ακολουθήσει ότι αν υπάρχουν τροπολογίες οι οποίες είναι μεταξύ τους ασύμβατες ή οδηγούν σε σύγκρουση με άλλα στοιχεία του κειμένου, εάν δεν είναι απαραίτητα όλα αυτά τα στοιχεία για να βελτιωθούν την σωστή ε, πορεία της έκθεσης, πιστεύω ότι θα πρέπει να μην γίνουν δεκτές. Μπορεί να έχουν σημασία και να είναι επίμαχες στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να διατηρήσουμε μέχρι ότου υπάρξει μια τελική απόφαση στην Επιτροπή μας. Επομένως αύριο εγώ θα καλέσω όλους αυτούς που συνέταξαν τροπολογίες σε μια συνάντηση, θα τους αποστείλω και προτάσεις συμβαστικών λύσεων και την εκτίμησή μου για τις δικές τροπολογίες και όπως είπε και ο κύριος ε, Μαργκάγιο και ο Ρωμάνος σοσιαλιστής ε, συντονιστής, όλα αυτά είναι ένα κοινό έργο στο οποίο πρέπει να αποδειθούμε όλοι και ελπίζω ότι με όλα αυτά θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια ευρεία συμφωνία και συνένεση για αυτό το τμήμα της, ε, του εποπτικού πακέτου. Κύριε Μπάλτς, θέλετε να λάβετε το λόγο μετά από όλα αυτά ή περιμένετε να έρθει το δικό σας κομμάτι του πακέτου. Ίσως είναι κάπως ε, άδικο να υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός μεταξύ των διαφορών αυτών κομματιών του πακέτου. Τώρα, θα δώσω το λόγο σε αυτούς που ζήτησαν το λόγο και ελπίζω ότι μπορούμε να περάσουμε τον περισσότερο χρόνο μας ακούγοντας τις απόψεις και από τα άλλα μέλη της Επιτροπής μας, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θέλετε να πείτε κάτι. Θα ήθελα απλώ να ξέρω πότε θέλετε να λάβω το λόγο και πάλι στο, θέμα αυτό. Ωραία λέει η πρόεδρος. Οι σκιώδεις εισηγητέ που θέλουν να λάβουν το λόγο μπορείτε να μας το πείτε και αυτό γιατί προς το παρόν έχουμε περίπου 27 άτομα που θέλουν να λάβουν το λόγο θα πρέπει να καταγράψουμε τα ονόματα και να καθορίσουμε ποιο χρόνο, πόσο χρόνο θα έχουμε στη διάθεσή μας. Εγώ θέλω να δώσω το λόγο πρώτα στους σκιώδεις εισηγητές και δίνω καταρχήν το λόγο στην Άστρεν Λούλινγκ γιατί ξέρω ότι είσαι σκιώδης εισηγήτρια Λούλινγκ και θα ήθελες να λάβεις το λόγο για το τραπεζικό τομέα, δεν κάνω λάθος. Ναι κυρία Πρόεδρε, είμαι σκιώδης για την έκθεση Γκουλάρ. Θα ήθελα δε να κάνω ένα σχολιάκι για, για την έκθεση του κυρίου Μαργκάλιου. Στο Financial Times ένα ενδιαφέρον άρθρο την περασμένη εβδομάδα ζητούσε να δημιουργηθεί μία αρχή επίλυσης διαφορών με τράπεζες. Θα ήθελα λοιπόν να μάθω γιατί δεν ζητάμε και εμείς τη δημιουργία ενός ουδέτερου οργανισμού που να διευθετεί τις διαφορές μεταξύ εθνικών αρχών για τα τραπεζικά. Νομίζω ότι θα ήταν πολύ πιο κομψό να δώσουμε μια τέτοια διαιτησία σε έναν ουδέτερο οργανισμό αντί να χρειάζεται ψηφοφορία για οριστική απόφαση Νομίζω ότι αυτά είναι περίεργα πράγματα. Ως προς τον τρόπο βέβαια εφαρμογής αυτής της ψηφοφορίας έχω καταθέσει μια τροπολογία ώστε να υπάρχει απλή πλειοψηφία. Έστω και με εξαιρέσει περισσότερο ή λιγότερο ευρείες. Καλύτερο αυτό παρά η προσφυγή συστηματικά στην ενισχυμένη πλειοψηφία που υπερπολιτικοποιεί τεχνικά απλώς θέματα. Ευχαριστώ λοιπόν τον κύριο Μαργκάλιο για αυτό το, αυτή την πρόταση και ελπίζω να τη δεχτούν και οι υπόλοιποι. Τώρα για την έκθεση Γκουλάρ που είμαι σκιώδης. Στην ομάδα μου εχθές κάναμε μια πρώτη εξέταση των συμβιβαστικών τροπολογιών που μας υπέβαλε η κυρία Γκουλάρ την περασμένη εβδομάδα και που συζητήθηκαν στο Στρασβούργο και επί των αρχών θα ήθελα να σας πω ότι η ομάδα μου υποστηρίζει τη θέση ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πρέπει να παίζει τον κυρίαρχο ρόλο στα πλαίσια της ΕΑΣΒΑ για τον απλό λόγο ότι είναι η πιο ευρωπαϊκή λύση αυτή διότι συμφωνεί με αυτά που προβλέπει η έκθεση Ντελαροζιέρ που κατανέμει ρόλους μεταξύ μακροεποπτείας και μικροεποπτείας που η τελευταία παραμένει δικαιοδοσία των εθνικών εποπτών. Η δε λογική του ανοίγματο που έχει τελικά υπερισχύσει καταλήγει να αμφισβητεί τον κυρίαρχο ρόλο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας πρέπει να ζητήσουμε τη γνώμη και άλλων εμπειρογνωμόνων και του κανονικού κόσμου κλπ. Γιατί όχι δεν είμαι κατά αλλά μέχρι τώρα εξάλλου έχουμε επιδείξει καλή θέληση. Τώρα όμως τίθεται το θέμα του μέχρι ποιο βαθμό θα ξεπεράσουμε τα προβλεπόμενα. Από πότε δηλαδή θα, θα παίζουν τόσο κυρίαρχο ρόλο οι εθνικές τράπεζες ώστε οι κεντρικές να μην, είναι πια, να μην έχουν πια τον πρώτο λόγο. Όσοι θέλουν τέτοιες διευρύνσεις νομίζω ότι θα καταλήξουν τελικά στην καταστροφή του ρόλου των κεντρικών τραπεζών. Εδώ δεν είναι αγώνας για θέσεις, αλλά το θέμα είναι όχι να δημιουργηθεί μια, ένας νέος οργανισμός που να ανταγωνίζεται ή συναγωνίζεται την ΕΚΤ, αλλά να είναι συμπληρωματικός ο ρόλος. Ό,τι και να γίνει θα παραμείνει η εποπτεία κατακαιρματισμένη και δεν χρειάζεται ένα νέο κυρίαρχο όργανο εφόσον η πραγματικότητα είναι κατακαιρματισμένη. Η εισηγήτρια κυρία Γκουλάρ λοιπόν τηρεί μια ενδιάμεση στάση. Η ΕΚΤ έχει αποδυναμωθεί σε σχέση με τους αρχικούς της στόχους. Η ιδέα αποδυνάμωση αυτή ζητούν οι σοσιαλιστές και οι πράσινοι να είναι ακόμη πιο μεγάλοι. Παράδειγμα, η Προεδρία ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας θα συμμετέχει και στην ΕΑΣΜΠ και ο αντιπρόεδρος αλλά θα προέρχεται εκτός Ευρωζώνης. Και ο δεύτερος αντιπρόεδρος τώρα, αν είναι εθνικός επόπτης ή ανήκει σε μία από τις τρεις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές, τότε θα υπάρχει κάποια εξισορρόπηση. Απ' την άλλη όμως υπάρχει ένα πρόβλημα. Ο πρόεδρος της ΕΑΣΜΠ θα βρίσκεται σε μειονοτική θέση μπροστά στο μέλος εκτός Ευρωζώνης και τον Εθνικό Επόπτη. Και απ' την άλλη αν λείπει θα αντικαθίσταται από έναν από τους αντιπροέδρους. Η Ευρωζώνη τότε μπορεί να μην εκπροσωπηθεί καθόλου. Και αυτό είναι προβληματικό. Γι' αυτόν τον λόγο τελικά προτείνω και οι δύο αντιπρόεδροι να είναι από την Ευρωζώνη. Θα μπορούσα επίσης να μιλήσω και για την ε, προσωρινή steering committee όπου πρέπει επίσης να υπάρχει μία εξισορρόπηση, δηλαδή δηλαδή να μην τροποποιηθεί η αρχική ισορροπία που, στην οποία βασίζεται το κείμενο αυτό αλλά και άλλα που αφορούν την ευρωπαϊκή εποπτεία. Τέλος κυρία Πρόεδρε θα καταθέσω ορισμένες συμβιβαστικές τροπολογίες ή μάλλον ορισμένες τροπολογίες προς τους συμβιβασμούς που προτείνει η κυρία Γκουλάρ και η ομάδα μου κατά τα άλλα νομίζω ότι είναι αρκετά μεγάλη ώστε να ε, ακουστούν αυτά που θα πούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Θα σας πω ποιοι άλλοι έχουν εγγραφεί για να μιλήσουν με τη σειρά με την οποία ζήτησαν το λόγο. Uh, Uh, and Sven Giegold, and then uh, from non-shadow. Και μετά από τους μη σκιώδεις, who... η Άννα Κοντζούρη. Αν θέλει κανείς άλλος να εγγραφεί. Τώρα λοιπόν ο κύριος Πιτέλας. Εγώ πιστεύω ότι το γενικό πλαίσιο που έχει παρουσιάσει ο κύριος Μαργκάγιο είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το δεχτούμε σε γενικές γραμμές. Για τους τρεις αυτούς κανονισμούς έχουμε ουσιαστικά για πρώτη φορά την απάντηση που μπορεί να δώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην κρίση των χρηματοπιστωτικών φορέων. Είναι απαραίτητο να εξασφαλίσουμε την εποπτεία των αγορών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οτιδήποτε άλλο σημαίνει ότι προδίδουμε τον ίδιο το στόχο της μεταρρύθμισης που είναι να δώσουμε μια απάντηση στις προσδοκίες πολλών πολιτών που έχουν θυγεί από την κρίση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μπορεί να αποσύσει την ευθύνη να αντιμετωπίσει τις προσδοκίες των πολιτών μονάχα και μόνο για να μπορέσει να υπάρξει μια συμφωνία με το Συμβούλιο. Δεν μπορούμε να θυσιάσουμε λοιπόν τους στόχους μας στην επίτευξη μιας σύντομης επίτευξης λύσης. Είναι απαραίτητο να εξασφαλίσουμε τους φορείς να έχουμε πραγματικά την ε, εποπτεία της ευρωπαϊκής αγοράς. Δεν μπορούμε να δεχτούμε να μην μπορούν αυτοί οι παράγοντες να παρεμβαίνουν στην αγορά. Ούτε μπορούμε να εξασφαλίσουμε την ε, εποπτεία χωρίς τη δυνατότητα να ανατρέπονται αποφάσεις που λαμβάνουν από εθνικούς ρυθμιστές. Αυτό θα ήταν λοιπόν μια λανθασμένη αντιμετώπιση μια αρνητική υπηρεσία στην Ευρώπη και δεν θα εξυπηρετούσαμε το στόχο της μεταρρύθμισης που να υπάρχει μια υπερεθνική εποπτεία. Για το άρθρο 10. Νομίζω ότι είναι απαραίτητο να έχουμε μια φιλόδοξη λύση και να απορρίψουμε άλλες απόψεις όπως το να δώσουμε στο Συμβούλιο την εξουσία να αποφασίζει πότε βρισκόμαστε ή πότε δεν βρισκόμαστε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Μια καλύτερη λύση και πιο λογική είναι να είναι ένα τεχνικό όργανο το οποίο θα αποφασίζει για κάτι τέτοιο και γι' αυτό υποστηρίζω τη θέση του κυρίου Γκίγκολτ, ο οποίο λέει ότι θα πρέπει να είναι το MSB, το Ευρωπαϊκό Συστη... Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου. Επίση πρέπει να είναι απαραίτητο να μπορεί να υπάρχει πρωτοβουλία της ε, Ευρωπαϊκής Αρχής για να επιλύει διαφορές μεταξύ ε, διαφορών εθνικών φορέων. Νομίζω ότι είναι απαραίτητο να τονίσουμε το ρόλο των, ε, ε, της ομάδας των ρυθμιστών για τα ιδρύματα που έχουν διαμεθοριακή λειτουργία. Είναι απαραίτητο λοιπόν να έχουμε και τους μηχανισμούς με τους οποίους θα έχει την εξουσία να το πράξει αυτό. Γι' αυτό στην τροπολογία μου προβλέπω να έχουν την υποχρέωση οι χώρες μέλη να κάνουν μια έκθεση αντικτύπου όταν ζητούν να γίνει δεκτό ότι μια δράση ρυθμιστικής αρχής έχει ε, επίπτωση στον προϋπολογισμό τους. Και έτσι μπορούμε να εξασφαλίσουμε μεγαλύτερη ασφάλεια για τους διάφορους τομείς. Νομίζω ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει και η δημιουργία ενός, ενός ε, ταμείου που θα αντιμετωπίζει την κρίση και που θα, δίνει, θα βασίζεται από τις εθνικές ε, συμμετοχές και αυτό θα μπορεί να αντιμετωπίσει τις μελλοντικέ κρίσεις. Και γενικά αποδέχομαι όλα αυτά τα οποία είπαν διάφοροι συνάδελφοι ότι θα πρέπει όλες αυτές οι αρχές να βρίσκονται σε μία μονάχα πόλη της Ευρώπης. Δεν θέλουμε εμείς να ακολουθηθεί το παράδειγμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιου με τις πολλές έδρες που είναι σε βάρος των πολιτών. Θέλουμε να έχουμε κάτι, να έχουμε κάτι το οποίο θα είναι κατανοητό και για τους εκλογείς μας και γενικά για τους φορολογούμενους στην Ευρώπη. Ευχαριστώ η Επανέρχομαι στην αρχή τη συζήτηση. Η δομή που συζητάμε υποτίθεται ότι θα προωθήσει τη σταθερότητα και τη διαφάνεια στον δημοσιονομικό τομέα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Κοινοί κανόνες και καλύτερη συνεργασία έτσι ώστε να διασφαλίζεται η εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου παντού και σε κατεπίγουσες περιπτώσεις και να εξυπηρετούνται ταυτόχρονα και τα συμφέροντα των φορολογουμένων. Αυτά είναι τα θετικά. Ξέρω ότι λόγω του σεισμού χάσαμε μια εβδομάδα, αλλά το κοινοβούλιο υποτίθεται ότι είναι δημοκρατικό και διαφανές. Ξέρω ότι οι συντονιστές και οι εισηγητές έκαναν πολλή δουλειά, αλλά για όποιον δεν είναι εισηγητής φοβάμαι ότι η συζήτηση υπήρξε, δεν υπήρξε καθόλου διαφανής και ίσως να είναι και χαοτική τολμώ να πω. Μπορούμε βέβαια να υποβάλουμε τροπολογίες. Και έχουμε τώρα και μια νέα έκδοση της έκθεσης με νέες τροπολογίες που συζητάμε σήμερα. Την επόμενη εβδομάδα θα ψηφίσουμε ίσως και με άλλες τροπολογίες που δεν τις ξέρει ακόμη κανείς. Πρέπει λοιπόν να είμαστε βέβαιοι ότι θα υπάρξει διαφάνεια και σε αυτή την επιτροπή και σε άλλες υπήρξε καλή συνεργασία μεταξύ εισηγητών και σκιωδών και ελπίζω το ίδιο να γίνει και με το έγγραφο αυτό. Υπάρχουν και μερικά νομικά όσο και πρακτικά προβλήματα για τις δικαιοδοσίες του οργανισμού αυτού. Στην αρχή έλεγαν οι να έχει ρόλο, να παίζει ρόλο εποπτείας άμεσα. Τώρα λένε να έχει χαρακτήρα υπηρεσίας, δηλαδή να τις μεταβιβάζονται εξουσίες από τις εθνικές αρχές. Και μόλις στις 15 Απριλίου υπόθηκε ότι δεν θα μπορεί να παίρνει αποφάσεις παρά μόνο όταν έχουν ταυτιστεί συγκεκριμένα τεχνικά προβλήματα χωρίς να έχει τον τελικό λόγο. Αυτό είναι πρόβλημα. Τι μου λέτε να μιλάω αργότερα, όχι, όχι. θέλει για διαδικαστικό να παρεύει κάποιος τώρα. Στο τέλος, τώρα, στο τέλος τώρα. Όχι στο τέλος. Εδώ για διαδικαστικό, αλλά στο τέλος. Ναι, καλά, εντάξει, ωραία. Συνέχισε, Βική, συνέχισε. Λοιπόν, χρειάζεται εδώ κάποιος χρόνος για να μπορέσουμε να επιδείξουμε διαφάνεια. Στην έκθεση Μαργκάλιο δεν γίνεται λόγος μόνο για ένα ταμείο αλλά για δύο πλέον. Και αυτό δεν έχει μπορέσει ακόμη να συζητηθεί. Εγώ το πήρα στις 5 παρα 10 χθες το δεύτερο αυτό ταμείο πρέπει να το εξετάσουμε. Έτσι ώστε να, γιατί προβλέπετε, να μπορεί να γίνει εγγύηση των καταθέσεων, χωρίς να ξέρουμε όμως αν θα πρόκειται για ένα σταθερό, μόνιμο, χρηματοπιστωτικό ίδουρημα. Ναι, εγώ δεν είμαι πεπισμένη ότι χρειάζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο τέτοια ίδρυμα. Όπως είπε και ο κύριος Σκίνερ, όλα αυτά τα θέματα να τα δούμε στα πλαίσια της έκθεσης Φεράρα με χρονοδιάγραμμα που να επιτρέπει όμως συζήτηση και για τους σκιώδεις. Μάλιστα, ο Ιωάννης Παύλος. Εγώ ήθελα να μιλήσω για δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα, είναι ένα θέμα στο που πρέπει να πω ότι παρίσταμε εδώ και πρέπει να λάβουμε υπόψη τις συστάσεις σας όσον αφορά το χρόνο αγόρευσης κυρίως όταν δεν έχουμε χρόνο στη διάθεσή μας. Επανειλημμένα ζητήσατε από τους παρεμβαίνοντες να είναι σύντομοι και δεν γίνονται πάντα σεβαστές αυτές οι προτάσεις για το χρόνο. Σας συντονιστής του ΕΛΚ και είναι ίδια άποψη έχουν άλλοι συντονιστές. Δεν θα πρέπει να είναι αδιαφανής αυτή η συζήτηση, να μην υπάρχουν πληροφορίες. Ποτέ στο Κοινοβούλιο στα έξι χρόνια που είμαι εδώ δεν είδα τέτοια συνεργασία μεταξύ συγγητών. Τέτοια συνεργασία μεταξύ των σκιωδών. Και η δουλειά που έκαναν οι συνάδελφοι, ε, οι συγγητές είναι πάρα πολύ σημαντική. Υπήρξαν ανοιχτοί, υπήρχε σωστή ε, μετάδοση των πληροφοριών. Είναι σημαντικό το έργο αυτό. Το χαρτοφυλάκιο είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την Ευρώπη δεν θα πρέπει να υποθεί ότι δεν εργάζεται διαφανώ το Κοινοβούλιο. Δεν υπάρχουν πολλοί θεσμοί στην Ευρώπη που εργάζονται με τέτοια διαφάνεια. Στη χώρα μου, οι συνεδριάσει των επιτροπών δεν είναι δημόσιε. Εδώ είναι δημόσιε. Δεν θα πρέπει να μιλάει κανεί άσχημα για τον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε εδώ σε αυτό το Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Θα πω κάποια λόγια στο τέλος, αν υπάρξει χρόνος, για την μεθοδολογία και άλλα συναφή. Διότι είναι πάρα πολύ δύσκολο το θέμα αυτό και το πακέτο. Ο Μάρκους Φέρμπερ είναι επόμενος στο κατάλογο. Ε, Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Είμαι σκιώδης εισηγητής για την οδηγία όμνιμους. Κάποιες παρατηρήσεις θέλω να κάνω. Πρώτα απ' όλα θέλω να διαπιστώσω ότι υπάρξει μια ανισότητα κάπως στην ποιότητα των ε, εκθέσεων στις οποίες έχουμε αντιμετωπίσει. Εγώ έχω δει με μεγάλη προσοχή αυτή την οδηγία και υπάρχουν, μάλλον η Κομισιόν, η Κομισιόν έχει επεξεργαστεί με έναν τρόπο άνισο την οδηγία γιατί το βλέπω αυτό στα σημεία τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσω ως και ο και πολλές φορές αυτό αφορά τεχνικά σημεία, σημεία που έχουν να κάνουν με την ε, προσαρμογή στη συνθήκη της Λισαβόνας και σημεία που έχουν να κάνουν με τους φόρους που πρέπει να δημιουργηθούν για το πακέτο εποπτείας δεν είναι πάντα εξαίρετο το έργο της Κομισιόν. Η Κομισιόν θα μπορούσε να είναι πολύ καλύτερη στην ε, επεξεργασία της στα σημεία αυτά. Δεύτερον θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή μου γιατί έχει κάνει μια πολύ, μια πολύ πλήρη παρουσίαση και καταφέραμε οι σχεδόν εισηγητές να καταλάβουμε λιγάκι καλύτερα για το ποια είναι η άποψή του για τις διάφορες τροπολογίες που έχει να αντιμετωπίσει. Ελπίζω ότι στη συνέχεια θα είναι πιο ευκρινής η άποψή του για όλα αυτά τα θέματα. Τώρα για το συνολικό πακέτο ήταν γνωστό ως πακέτο λαμφαλουσής στις προηγούμενες θητείες του Κοινοβουλίου και υπάρχει το πραγματικό ερώτημα του πώς θα μπορέσει να αντιμετωπιστεί αυτό μέσα στη νέα δομή επιτροπολογίας που θεσπίζει η συνθήκη της Λισαβόνας για τις καθεξιοδότηση πράξεις Εδώ θα πρέπει να εξασφαλίσουμε την ε, συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως προβλέπουν λοιπόν οι συνθήκες και εδώ θα ήμουν ευγνώμων αν ακολουθήσουμε μια πιο σόφρονα διαδικασία και δεν μπορούμε να έχουμε μια βεβαιασμένη διαδικασία. Ο εισηγητής προβλέπει έξι μήνες για να προχωρήσει αυτή η διαδικασία και να είμαστε σε θέση να προχωρήσουμε μαζί με τις ε, συμβουλευτικές επιτροπές για να καταλήξουμε σε κάποιο συμπέρασμα. Και όχι μονάχα τρεις διαδικασίες, τρεις μήνες όπως η διαδικασία Λαμφαλουσί. Ανέφερα όμως για ορισμένα θέματα ότι τέσσερις μήνες θα ήταν επαρκής. Θα ήθελα να έχω λοιπόν μια σαφέστερη άποψη για τον συγητή γιατί και εγώ έχω πολλούς, πολλές αμφιβολίες για μια διαδικασία η οποία θα είναι ταχεία διαδικασία. Πρέπει να έχουμε μια λογική διαδικασία. Το να έχουμε μόνο τροπολογίες δεν σημαίνει ότι θα υπάρξει και ουσιαστική τροποποίηση του νομοθετήματος. Μια άλλη παρατήρηση. Φαίνεται ότι τα καταφέραμε να έχουμε κάποια συνένεση η οποία ξεπερνάει τα στενά κομματικά πλαίσια αλλά θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει και με το Συμβούλιο, πώς θα αντιμετωπίσουμε την πρόκληση μιας συμφωνίας με το, με Συμβούλιο. Αν δεν έχουμε μια συνεκτική αντιμετώπιση σε σχέση με τις επιμέρους ε, οδηγίες και τις ε, επιμέρους αρχές οι οποίες θα πρέπει να θεσπιστούν, θα έχουμε πολλές δυσκολίες με το Συμβούλιο, γιατί το Συμβούλιο έχει ουσιαστικά αποφασίσει ομόφωνα για τα θέματα αυτά. Αυτή τη στιγμή οι αγορές και ο χρηματοπιστωτικός τομέας δεν πλήττεται από υπερβολική Ευρώπη, αλλά υπερβολικό αριθμό απόψεων των κρατών μελών, που είναι διαφορετικές. και ίσω η Ευρώπη αυτή τη στιγμή δεν είναι υπερβολικά μεγάλη, αλλά ίσω είναι υπερβολικά μικρή για να μπορέσει να επιβάλλει κανόνε συνεκτικού στον τομέα τη αγορά. Αλλά προφανώ τα κράτη-μέλη δεν μπορούν να το κάνουν μεμονωμένα. Γι' αυτό πιστεύω ότι στο συμφέρον των πολιτών, των επενδυτών στην Ευρώπη, θα πρέπει εμεί να κάνουμε μια προσπάθεια να καταλήξουμε σε μια κυρίω συνεκτική στάση για τα θέματα αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστώ. Άντωνη, θε να αναφερθεί σε κάτι άλλο. Eh, Ευχαριστώ, λέει ο κύριο Σάντσε Πεσέδο. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Γκαρσία Μαργάγιο για τη δυνατότητα που μα έδωσε να έχουμε μια στενή επαφή μαζί του όλο αυτό το διάστημα και να μιλήσουμε επί της ουσίας για όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την εποπτεία των τραπεζικών ε, φορέων. Βέβαια δεν μπορούμε να επιλύσουμε μέσα σε μια μικρή συζήτηση όλο αυτό το πολύπλοκο θέμα και μέχρι τη στιγμή που θα υπάρξει οριστική απόφαση από την Ολομέλεια παραμένουν πολλά θέματα εκκρεμή. Όχι μονάχα για λόγου χρονοδιαγράμματο, αλλά και αυτοί παίζουν κάποιο ρόλο. Ξεκινήσαμε το τελευταίο τρίμηνο του 2009 την εργασία μα και πιστεύω ότι θα πρέπει να τελειώσουμε με κάποια οκίτητα την εξέταση αυτού του θέματο. Η απόψη μου είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ω παγκόσμιο ηγέτη στον τομέα των τραπεζών και τον τομέα των ασφαλιών θα πρέπει να έχει κάποιες προτάσεις για την επόμενη σύνοδο των G20 το 26-27 Ιουνίου για να μπορέσει να παίξει κάποιο καθοριστικό ρόλο στη διαδικασία μεταρρύθμισης στον τραπεζικό και ασφαλιστικό τομέα. Αλλά υπάρχουν πολλά θέματα για τα οποία πρέπει να προχωρήσουμε σε σημαντικές συζητήσεις και ίσως θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας στις πτυχές αυτές όπου νομίζουμε ότι υπάρχει μια επαρκής ορίμανση για να καταλήξουμε σε μια κοινή στάση από την πλευρά της Ευρώπης. Χωρίς φυσικά αυτό να είναι εξαντλητικό. Δεν μπορούμε <clears throat> να θεωρήσουμε ότι έχουμε επιλύσει πάρα πολλά από τα προβλήματα τα οποία απαιτούν ακόμα πιο ενδελεχή αντιμετώπιση. Πιστεύω ότι όσο έτσι που προχωρούν τα θέματα αυτά είναι η δεύτερη μονάχα φορά που συζητούμε τις τροπολογίες έχει δημιουργηθεί μια κρίσιμη μάζα που μπορεί να μας επιτρέψει να καταλήξουμε σε μια συνεκτική στάση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο σημείο αυτό. Ακόμα και αυτοί που συμφωνούν δεν είναι σίγουροι με τον εαυτό τους ότι συμφωνούν σε όλα αυτά τα στοιχεία. Πιστεύω ότι υπάρχει ένα υψηλό επίπεδο συνένεση και πρόκειται για μια διαδικασία η οποία έχει εκμεταλλευτεί τις διάφορες προτάσεις από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, από την Κομισιόν, από την Επιτροπή Λαρόσια. Ξέρουμε και ποιε είναι οι του Συμβουλίου και πιστεύω ότι οι βασικές ε, συμφωνίες που επέτυχε η Σουηδική Προεδρία από το Συμβούλιο ήταν κάπως ανεπαρκής και γι' αυτό θα πρέπει να προχωρήσουμε επέκεινα αυτών. Τα σημεία τα οποία για μένα είναι τα πιο σημαντικά και στα οποία έχει υπάρξει κάποια πρόοδο σε ορισμένε πτυχές Καταρχήν το θέμα της ε, βιωσιμότητας σε χρηματοοικονομικό επίπεδο δεν αναφέρεται αυτό εκπεφρασμένα, αλλά αναφέρεται η ανάγκη να διατηρήσουμε μια σταθερότητα, η οποία δεν πρέπει να είναι μόνο βραχυπρόθεσμη, αλλά πρέπει να είναι και μακροπρόθεσμη. Είναι σημαντικό λοιπόν αυτό το θέμα της σταθερότητας. Δεν θέλουμε να περιοριστούμε μονάχα σε ρητορικέ δηλώσεις. Τονίζουμε την ανάγκη να υπάρξει σωστή διάδραση μεταξύ του χρηματοοικονομικού τομέα και του τομέα της πραγματικής οικονομίας. Επίσης να εξασφαλίσουμε το θεμητό ανταγωνισμό. Αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα. Και, το δεύτερο, και επίσης επιπλέον το θέμα της ενσωμάτωσης του, του εξωτερικού κόστους. Για όλα αυτά τα θέματα υπάρχει επαρκής πιστεύω βαθμός συνένεσης. Ένα άλλο θέμα είναι το πώς θα μπορέσουμε να έχουμε μια εποπτεία η οποία δεν θα είναι απλώς τεχνική αλλά θα έχει και προληπτικό χαρακτήρα. Και εδώ πιστεύω ότι είναι απαραίτητο να έχουμε μια μορφή εποπτείας που προσθέτει αξία σε σχέση με την ίδια υπάρχουσα εποπτεία που αφορά κυρίως τα θέματα κίνδυνου. Εμείς θελήσαμε να υπάρξει ένας καλύτερος ορισμός του συστημικού κινδύνου και του διαμεθοριακού κινδύνου ή να έχουμε ένα ορισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο που σε ό,τι αφορά τους κινδύνους να περιλαμβάνει και τους διαμεθοριακούς κινδύνους. Εγώ είμαι έτοιμο να δεχτώ μια τέτοια διατύπωση σε θεολογικές σκέψεις και να προχωρήσω περισσότερο. Και ιδίω θα πρέπει να δούμε πώς θα γίνει αυτή η πολυεπίπεδη μορφή εποπτείας, δηλαδή πώς θα μπορέσει να λειτουργήσει η ευρωπαϊκή εποπτεία μαζί με τις εθνικές μορφές εποπτείας. Είναι απαραίτητο να έχει ένα οριζόντιο χαρακτήρα η ευρωπαϊκή εποπτεία αυτό είναι κάτι το οποίο τονίστηκε σε όλε τι συζητήσει, Αν θέλουμε να έχει συνεκτικό χαρακτήρα αυτή η εποπτεία και να υπάρχει ο ενιαίος, το ενιαίο σύνολο κανόνων, το single rule book όπω λέμε, δεν μπορεί να υπάρχει ένας σύνολο κανόνων για ορισμένου φορεί και ένας άλλος για όλου του τομείς. Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει μια ευρωπαϊκή εποπτεία με ενιαίο βιβλίο κανόνων. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι κανόνες για τους ε, κινδύνους θα πρέπει να εφαρμόζονται με απόλυτα μηχανιστικό τρόπο. Θα πρέπει να υπάρχει για όλους τους συστημικούς φορείς ενιαίοι κανόνες οι οποίοι δεν θα τροποποιούνται. Μπορούν οι κανόνες να διαμορφώνονται σε σχέση με τους κινδύνους, αλλά οι κανόνες για την εκτίμηση του κινδύνου θα πρέπει να είναι ήδη. Λοιπόν, να προσθέσουμε και κανόνες όταν αυξάνεται ο κίνδυνος, αλλά αυτοί οι κανόνες θα πρέπει να διαμορφώνεται σε σχέση με το κίνδυνο και όχι σε σχέση με διαφορετική φύση φορέων. Αυτό νομίζω ότι είναι απαραίτητο. Για να υπάρχουν αποτελεσματικοί κανόνες, εμείς θα πρέπει να θεσπίσουμε και τον κατάλογο των εξουσιών και να εξασφαλίσουμε μια μεγαλύτερη ομοιογένεια. Γιατί οι αρχές, οι ρυθμιστικές θα πρέπει να είναι αυτές οι οποίες θα εξασφαλίσουν τη σωστή εφαρμογή των ευρωπαϊκών οδηγιών. Αν όλες αυτές εφαρμόσουν την ίδια οδηγία θα πρέπει να έχουν ισοδύναμες εξουσίες. Αυτό είναι κάτι το οποίο παραμένει ακόμα εκρεμές και δεν έχει επιληθεί. Πρέπει να έχουν την ισχύ να εφαρμόσουν αυτές τις οδηγίες και αυτό αναφέρεται και στα τεχνικά πρότυπα. Τα τεχνικά πρότυπα θα πρέπει να αντιμετωπιστούν κυρίως με κάτι εξουσιοδότηση πράξης της Κομισιόν, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει μια πιο στεναρή μνήα στο ενιαίο βιβλίο κανόνων και θα επιμείνουμε εκεί ως το τέλος. Επίσης, να πρέπει να εξασφαλίσουμε μια μεγαλύτερη ανεξαρτησία των εποπτικών αρχών. Και αυτό έχει να κάνει και με τα θέματα του προϋπολογισμού. Εδώ έχουμε να αντιμετωπίσουμε λοιπόν αυτό το πολύ σημαντικό πρόβλημα και επίσης σε ό,τι αφορά το ότι πρέπει να έχει συμμετοχικό χαρακτήρα η εποπτεία με ευρεία συμμετοχή σε συμβουλευτικό τουλάχιστον επίπεδο. Αυτό προσπαθούμε λοιπόν να προωθήσουμε και είναι απαραίτητο σε δημοκρατικό επίπεδο για να συμπεριληφθεί και ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Υπάρχει και μια ακόμα πτυχή που νομίζω ότι προς το παρόν δεν έχουμε προωθήσει ιδιαίτερα. Δεν αναφέρομαι στην εποπτεία των συστημικών φορέων, αλλά στη συστημική εποπτεία. Είναι μια ευρύτερη έννοια αυτή. Θα ήταν δηλαδή χρήσιμο να ξέρουμε τι ακριβώς αποτελεί το συστημικός κίνδυνος, πώς μπορούμε να ανοιχνεύσουμε τον συστημικό κίνδυνο και να βρούμε αυτές τις δραστηριότητες οι οποίες επέχουν συστημικούς κινδύνους και να δούμε στη συνέχεια ποια είναι τα εργαλεία τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας και ποια είναι τα δίκτυα ασφαλείας τα οποία θα πρέπει να θεσπίσουμε. Είναι απαραίτητο να τονίσουμε ότι η πρώτη μας προτεραιότητα θα πρέπει να είναι η προστασία των καταθετών και δεύτερον η ενσωμάτωση όλων των πηγών κόστους και τέλος δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ήδη μια κρίσιμη μάζα, δεν χρειάζεται να αναβάλουμε στο δυναμικές τις αποφάσεις. Βρισκόμαστε ήδη σε μια διαδικασία όπου θα πρέπει να κάνουμε κάποια βήματα και να τροποποιούμε την ε, στάση μας στην πορεία, διότι είναι μια διαδικασία που δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι έχει κλείσει ακόμα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να τονίσω την ε, ανάγκη να ευθυγραμμίσουμε τις τρεις αυτές από τις εκθέσεις και αυτήν φυσικά για τις ασφάλειες και τις συντάξεις την οποία είμαι σχεδόν εισηγητής. Θέλω να, θεωρήσω, να τονίσω ότι είναι απαραίτητο το άρθρο 2 της έκθεσης για τις ασφάλειες να ευθυγραμμιστεί με τις άλλες έκθεσεις. Υπάρχουν ασφαλιστικοί φορείς οι οποίοι παρουσιάζουν και αυτοί ένα συστημικό χαρακτήρα. Αυτό το τόνισε η Ένωση των Ασφαλιστικών Φορέων στην Γενέβη στην έκθεσή της. Και επίσης υπάρχουν κανόνες που αφορούν τις τράπεζες οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν και στην περίπτωση των ασφαλιών. Να υπάρχει λοιπόν ένας, ένα ταμείο για τις ε, ασφάλειες. ένα τέτοιο, ένα τέτοιο ταμείο θα απαιτούσε πολύ λιγότερους πόρους από ό,τι στην περίπτωση ενός ταμείου για το τραπεζικό σύστημα. Επίσης γνωρίζουμε Ποιε είναι οι ιδιαιτερότητε του τομέα του ασφαλιστικού που κάνουν πιο απίθανες ή πιο σπάνιες τις πτωχεύσει στον τομέα αυτό. Επίσης, αντίθετα με τις τράπεζε, τα χαρτοφυλάκια των ασφαλιστικών εταιριών μπορούν να πάνε σε άλλους φορείς με συστήματα ασφάλεια και να ελαχιστοποιήσουν τις περιπτώσεις όπου χρειάζεται διάσωση ενό ασφαλιστικού φορέα. Προτείνουμε επίση να δημιουργηθεί ένας ευρωπαϊκό, ένα ευρωπαϊκό η Ευρωπαϊκή Τράπεζα για τα συστήματα εγγύησης των ασφαλιστικών τομέων, ώστε να μπορέσει αυτή η Ευρωπαϊκή Αρχή να έχει όλα τα συστήματα ασφάλισης των εθνικών ασφαλιστικών φορέων. Να υπάρχει ένα σύστημα τέτοιο για κάθε κράτος μέλος, να υπάρχει ένα επίπεδο κοινό σε όλους τους ε, εθνικούς φορείς σε ευρωπαϊκό επίπεδο και επίσης ένα σύστημα ασφαλείας για τους ασφαλιστικούς φορείς που παρουσιάζουν συστημικούς κίνδυνους. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Φέρμπερ. Κύριος Γκόρι τώρα έχει το λόγο. Κυρία Γκόρι. Έχω μία παρατήρηση νομίζω ότι θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας στα θέματα τα οποία είναι επίμαχα ή θα μπορούν να είναι επίμαχα, ιδίως στις συζητήσεις με το Συμβούλιο. και θα πρέπει να δούμε πώς θα μπορούσαμε να κινηθούμε για να καταλήξουμε σε μια συμβαστική λύση με το Συμβούλιο. Είναι απαραίτητο να εξασφαλίσουμε τη λειτουργία αυτών των εποπτικών αρχών το ταχύτερο δυνατό Ποια είναι ακόμα τα σημαντικά θέματα τα οποία έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Καταρχήν, οι αρμοδιότητες ε, σε επίπεδο αποφάσεων αυτών των αρχών οι οποίες θεσπίζονται. Το Κοινοβούλιο υποστηρίζει μια ευρωπαϊκή εποπτεία. Θα πρέπει να είναι υποχρεωμένες αυτές οι αρχές να αναλαμβάνουν τις αντίστοιχες ε, αποφάσεις που θα καλύπτουν τους φορείς ευρωπαϊκής συστημικής σημασίας. Εδώ θέλω να θέσω και το εξή ερώτημα στους εισηγητές. Σε πολλές χώρες υπάρχουν τράπεζες που ανήκουν σε ξένους. Όταν εμείς θέλουμε να έχουμε φορείς εποπτείες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πώς θα μπορέσει να λειτουργήσει στις τράπεζες αυτές. γιατί υπάρχουν αυτές οι τράπεζες που δεν έχουν ουσιαστικά ευρωπαϊκή ιδιοκτησία. Πώς θα λειτουργήσει λοιπόν αυτή η διαδικασία για να αντιμετωπιστεί και η αντίστοιχη ευθύνη αυτών των τραπεζικών φορέων. Μήπως υπάρχουν κίνδυνοι οι οποίοι συνδέονται με τις ε, χώρες αυτές όπου υπάρχουν τραπεζικά ιδρύματα τα οποία ελέγχονται από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μήπω στην περίπτωση που υπάρχουν Ευρωπαίοι επενδυτέ, θα πρέπει να εξασφαλίζεται και η εποπτεία από ευρωπαϊκούς φορεί. Και αν θα πρέπει να υπάρχει έλεγχος από την Ευρωπαϊκή Αρχή και όχι μονάχα από τις Εθνικές Αρχές. Επίσης θα πρέπει να εξασφαλίσουμε την παρουσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να έχει πάντα μία ψήφο στην διαδικασία αυτή της εποπτικές αρχές. Αυτό δεν είναι λοιπόν μονάχα ένα πολιτικό θέμα, αλλά και θέμα του να εξασφαλίσουμε την επαγγελματική επάρκεια αυτών οι οποίοι θα βρίσκονται στην εποπτική αρχή. Πιστεύουμε λοιπόν ότι να εφαρμοστεί η λειτουργία αυτών των εποπτικών αρχών με ένα σταδιακό τρόπο, ώστε να μην υπάρξει στρέβλωση ανταγωνισμού και να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρξουν και ζημίες στο σύστημα. Και επίσης το θέμα των τεχνικών προτύπων είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε στον τομέα αυτό οι ευρωπαϊκές αρχές εποπτικού χαρακτήρα να μην προχωρήσουν σε λεπτομέρειες για θέματα τα οποία δεν είναι παρά μόνο επουσιώδη. Μπορούμε λοιπόν να αφήσουμε το θέμα αυτό σε μεγάλο βαθμό στις εθνικές αρχές. Το επόμενο σημαντικό ερώτημα είναι το θέμα της εξασφάλισης ασφάλειας δικαίου για τα κράτη-μέλη. Ποιες θα είναι οι δυνατότητες για τα κράτη-μέλη όταν δεν συμφωνούν με μια συμφωνία της Ευρωπαϊκής ε, Εποπτικής Αρχής. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ζητήσει πάντα να υπάρχει μια έκθεση αντικτύπου εάν θέλουν τα κράτη-μέλη να αποδείξουν ότι υπάρχουν αρνητικές συνέπειες σε επίπεδο προϋπολογισμού. Αλλά ένα διάστημα 10 ημερών δεν μου φαίνεται επαρκής. Θα πρέπει τουλάχιστον να υπάρχει ένας μήνας στη διάθεσή τους. και για την ε, παροχή πληροφοριών. Είναι απαραίτητο να μπορούν να παίρνουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες οι αρχές εποπτείας, αλλά χωρίς τόσο μεγάλη λεπτομέρεια ώστε αυτό να αποβεί εις βάρος των χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων. Επίσης η σημασία, η συμμετοχή των κεντρικών τραπεζών στον, στους φορείς εποπτείας. Πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα να συμμετέχουν οι εθνικές κεντρικές τράπεζες στους φορείς εποπτείας γιατί έχουν τις δικές τους τράπεζες δεδομένων με τις οποίες μπορούν να παρακολουθήσουν τα θέματα ιδίως ρευστότητα και επομένως θα πρέπει να υπάρχει παρουσία τους. Μερικές καταληκτικές ε, παρατηρήσεις. Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να έχουμε μια συμβουλευτική τεχνική επιτροπή η οποία θα έχει ισχυρό ρόλο και θα περιλαμβάνει εμπειρογνώμονες από τις ε, κεντρικές τράπεζες για συγκεκριμένα θέματα τα οποία απαιτούν εμπειρογνωμοσύνη και υπήρξαν και προτάσεις να έχουμε και ακαδημαϊκούς ερευνητές ε, σε, αυτές τις, ε, σε αυτούς τους φορείς. Αυτό ίσως είναι υπερβολικό και για, επίσης για το, το Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου δεν είναι απαραίτητο εδώ να υπάρχουν εθνικοί εμπειρογνώμονες γιατί εδώ τίθενται κυρίως τομεακά θέματα. Μάλλον τίθενται γενικά και όχι τομεακά θέματα. Και επίσης πιστεύω ότι είναι απαραίτητο να υπάρξει εκπροσώπηση στη εποπτική αρχή εμπειρογνωμόνων αλλά δεν πρέπει να έχουν τον προσέρχοντα ρόλο σε αυτό το φορέα. Υπάρχουν επίσης πολλές τροπολογίες ώστε να συμμετέχουν και χώρες εκτός της ζώνης του ευρώ στην εποπτική αυτή αρχή και νομίζω ότι πρέπει ο κανονισμός να αναφέρει τη δυνατότητα εκπροσώψεις και των χωρών αυτών, γιατί όταν προκύπτουν κρίσεις δεν υπάρχει όριο στο οποίο περιορίζεται η κρίση, θα πρέπει και οι χώρες αυτές εκτός της ζώνης του ευρώ να μπορούν να συμμετέχουν. Πιστεύω λοιπόν ότι και αυτό το θέμα θα πρέπει να ρυθμιστεί. Καλώς, ο Σφέν. Μπορείς να ξαναπάρεις το λόγο και μετά εκεί και μετά εγώ. Πολύ σύντομα ως σκιώδης για το ESRB θα ήθελα να προσθέσω ότι σαν πράσινοι εξακολουθούμε να αντίχουμε πρόβλημα. Ξέρουμε ότι είμαστε μειοψηφία, αλλά θα ήθελα να πω ότι εξακολουθούμε να έχουμε πρόβλημα με τη λογική επαναλήψεως σε όλα τους θεσμούς. Τη λογική ότι 27 κράτη-μέλη πρέπει να εκπροσωπούνται στου φορεί λήψη αποφάσεων με του εκπροσώπου των κεντρικών του τραπεζών. Πρέπει να πω ότι υπάρχει κάποια διαφορά μεταξύ τη λογική αυτής τη λογικής που έθεσε η κυρία Λούλινγκ που έλεγε ότι θέλουμε ευρωπαϊκή λύση. Αυτό από τη μια και από την άλλη να μην μπορούμε να επιλέγουμε κάποιους ανθρώπους, αριθμό ανθρώπων που θα και να περιορίσουμε το μέγεθος των φορέων. Να μην υπάρχει υπερβολικός πλουραλισμός. Εγώ συμφωνώ ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα πρέπει να ηγείται του ESRB. Εκεί δεν υπάρχει διαφορά στην ε, Επιτροπή. Δεν υπάρχει απόκριση. Ευχαριστώ και... Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Είναι πολύ σημαντικό να πω ότι πολλά υπόθηκαν τώρα που ήρθα εγώ καθυστερημένα. Θέλω να επικεντρωθώ επί της διαδικασίας από εδώ και πέρα. Ο Ζαν Πολ έκανε κάποια σχόλια, εγώ θα είμαι όσο πιο σύντομη γίνεται. Εγώ ήμουν ασκιώδης για το έγγραφο περιασφαλίσεων και παρόλο που κατάφερα να φτάσω την πεσμένη εβδομάδα στο Στρασβούργο και να απολαύσω τη λιακάδα, δεν μπόρεσα να μιμηθούν πολύ και χάσαμε μια ολόκληρη εβδομάδα που είχαν προγραμματιστεί πολλέ συναντήσει για το έγγραφο για τι ασφαλίσεις και χάσαμε πάρα πολύ χρόνο. Χάσαμε και αυτή την εβδομάδα για το έγγραφο για τι ασφαλίσει, διότι η παρόλο που δεν έφταιγε δεν είναι διαθέσιμο όλη την εβδομάδα. Χάνουμε δύο ολόκληρε εβδομάδε για το έγγραφο για τι ασφαλίσει σε πολύ κρίσιμη καμπή αν πρόκειται να ψηφίσουμε στις 4 Μαΐου. Υπάρχουν θέματα. Το έγγραφο τη ασφαλίσεως, όπως είπαν και πολλοί άλλοι, έχει διαφορετική μορφή σε σχέση με τα άλλα δύο. Και στόχος είναι να πλησιάσουμε τα έγγραφα όσο γίνεται περισσότερο και να παραμείνουν όσο πιο κοντά γίνεται. Και γι' αυτό έχουμε πάρα πολλή δουλειά να κάνουμε. Ε, ή να πλησιάσουμε τις δύο εκθέσεις κοντά στη μία ή τη μία κοντά στις άλλες δύο. Αλλά δεν είμαστε κοντά στη φάση όπου αυτά τα τρία έγγραφα είναι συγκρίσιμα ή ακολουθούν τις ίδιες ε, γραμμές όσον αφορά την αρχή σε τέσσερις εργάσιμες ψηφίζουμε. Δεν έχουμε διαθέσιμο εισηγητή για τρει από αυτέ τι μέρε για το έγγραφο τη ασφαλίση και ανησυχώ. Δεν είδα κατάλογο ψηφοφοριών που θα είναι πάρα πολύ περίπλοκοι, θα πρέπει να του επεξεργαστούμε. Πώ το καλό διαδικαστικά θα ψηφίσουμε στις 4 Μαΐου. Κανονικά θα τα έλεγα αυτά στη συνεδρία των συντονιστών που ανεβλήθη από την περασμένη εβδομάδα. Οπότε τώρα έχουμε συνεδρία συντονιστών για να αποφασίσει τη διαδικασία αφού γίνει η ανταλλαγή των απόψεων σήμερα τα πάντα είναι αντίστροφα και αναστατωμένα. Δεν φταίει αυτή η Επιτροπή. Έτσι συνέβησαν τα πράγματα. Ποια είναι η πραγματικότητα, όπως από τα πράγματα. Το πρόγραμμα της ΕΚΟΦΗΝ δεν έχει προγραμματίσει σύντομα την αρχιτεκτονική, την εποπτική. Άρα θα ήθελα να συμφωνήσω με τον Μπούλμαν. Να κάνουμε καλή δουλειά και να μην προχωρήσουμε γρήγορα και τελικά καταλήξουμε σε λάθος αποτέλεσμα. Θα πρέπει να συζητήσουμε τις τροπολογίες για όλα τα έγγραφα. Θα πρέπει να έχουμε το χρόνο να τις εξετάσουμε διεξοδικά. Οπότε αν δημιουργηθούν οι θεσμοί τον Ιανουάριο του 2011 να μην δημιουργηθούν πολλά προβλήματα. Νομίζω ότι θα πρέπει να εξετάσουμε τη διαδικασία μέσω της οποίας θα φτάσουμε εκεί και πώς θα το πετύχουμε σωστά αντί να τα στριμώξουμε όλα στις επόμενες τέσσερις ημέρες. Αυτό πρέπει να προσέξουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι βέβαιη ότι τα πράγματα θα διορθωθούν, αλλά είναι απαραίτητο να δούμε και το χρονοδιάγραμμα. Πάντοτε λέγαμε ότι θα προσπαθούσαμε να εργαστούμε το δυνατόν γρηγορότερα, χωρίς όμως να θυσιάσουμε την ποιότητα της δουλειάς μας. Και ισχύει αυτό. οι συντονιστές αργότερα σήμερα θα συζητήσουν αν μπορούμε να καθυστερήσουμε την ψηφοφορία χωρίς αυτό να διαταράξει τη λειτουργία του Κοινοβουλίου. Θα δούμε πώς λειτουργεί και ο τριμερής διάλογος Θα δούμε τι θα γίνει με την διαπραγματευτική ομάδα και σε τι επίπεδο θέλουμε να γίνει ο τριμερής. Αν θέλουμε να έχει ιδιαίτερα πολιτικό χαρακτήρα ή όχι. Αν θέλουμε να είναι υψηλού πολιτικού περιεχομένου. Όλα αυτά πρέπει να αποφασιστούν. Υπάρχουν και άλλα προβλήματα βέβαια, αλλά τα φροντίζουν. Η κυρία Σάντσες προσπαθεί να δει αν η πίεση που ασκεί το Κοινοβούλιο στο σύνολό του βολεύει και την Επιτροπή μας ή όχι. Επίσης, αύριο θα συναντήσω εκπροσώπους της Ισπανίας για να δούμε τι μεθοδολογία θα ακολουθήσουμε μετά την ψηφοφορία. Και μου λέει η γραμματεία ότι σήμερα το απόγευμα θα δούμε και το πρώτο σχέδιο της, ε, του καταλόγου των ψηφοφοριών. προσωρινός θα είναι βέβαια, αλλά θα δούμε το έστω το, την προσωρινή σειρά με την οποία θα ψηφιστούν οι τροπολογίες. Θα βοηθήσει και αυτό. Η ημερομηνία της ψηφοφορίας τώρα είναι κάτι που πρέπει να το ξαναδούμε γιατί αν υπάρξουν πολλές τροπολογίες μπορεί να μην μπορέσουμε να ψηφίσουμε στις 4 Μαΐου. Αλλά δεν θα το αποφασίσω εγώ όλοι μαζί, όλοι μαζί. Τώρα, αν θέλει κανείς να ξαναμιλήσει αλλά με την αντίθετη σειρά από την προηγούμενη. Διότι οι έσχατοι έσονται πρώτοι, έτσι έχει υποθεί. Αλλά και οι πρώτοι έσχατοι. Θέλει κανείς συντονιστή ή συντονίστρια, όχι. Ε, τότε εσύ. Συγγνώμη, αλλά πρέπει να επανέλθω συντόμως. Λοιπόν, το σημαντικό τώρα <clears throat> δεν είναι η ταχύτητα, αλλά ο τρόπος με τον οποίο θα λειτουργήσουμε. Έχουμε ένα υπεροκιάνιο το οποίο οδηγούμε και όταν πάρει μια κατεύθυνση είναι πολύ δύσκολο να αλλάξουμε πορεία σε ένα μεγάλο πλοίο. Γι' αυτό είναι σωστό και απαραίτητο να βρούμε τη σωστή κατεύθυνση. Φυσικά για μένα έχει μεγάλη σημασία από πατριωτική άποψη να εγκριθεί αυτό το έγγραφο υπό Ισπανική Προεδρία. Αλλά δεν είναι αυτό το ουσιώδες. Η προβληματική την οποία αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή έχει ένα προσωρινό χαρακτήρα. Θέλω να ευχαριστήσω τον Ζωάν Πολ Γκοζές για την υποστήριξη που έδωσε σε όλους τους εισηγητές. Έχουμε εργαστεί ουσιαστικά χωρίς τις τροπολογίες σε μεταφρασμένη μορφή εργαστήκαμε σε μια γλώσσα που δεν είναι δική μας και έχουμε διατηρήσει μια μόνιμη επαφή μεταξύ μας για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Το ερώτημα το οποίο ανέφερε και η εκπρόσωπος της συντηρητικής ομάδας είναι αν υπήρξε μια συμφωνία να διανεμηθούν οι εκθέσεις αυτές σε τέσσερις διαφορετικές ομάδες επί τη βάση της αρχικής τους <clears throat> φιλοσοφίας. Ιδίω για να βρούμε τεχνικού χαρακτήρα λύσεις. Το... Οι Βρετανοί συντηρητικοί χωρίσανε από την ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο και αυτό επηρεάζει τη σημερινή του κατάσταση, το αν είχαν μια έκθεση ή όχι. Εγώ παρόλα αυτά συμφωνώ με όλε τι πολιτικέ ομάδε ότι για να συζητήσουμε θα πρέπει να μπορέσουμε να φτάσουμε σε κοινέ απόψει μεταξύ ατόμων που έχουν κάποιο κοινό υπόβαθρο. Γι' αυτό προσπαθήσαμε να καταλήξουμε σε κάποιο εδρεωμένο, ενοποιημένο κείμενο και θα σας πληροφορούμε για το ποιε είναι οι προσωρινές μας συμφωνίες εν καιρό. Το βασικό θέμα τώρα είναι το θέμα <clears throat> του πώς θα γίνεται η εποπτεία του κινδύνου και ενδεχομένως των συστημικών φορέων. Η κυρία Γκουλάρ λέει ότι αυτό είναι πρόβλημα μόδας δεν είναι θέμα μόδας για μένα. Πολλές φορές βλέπετε ότι δεν έχει αλλάξει η απόψή μου επειδή περνάω από το φθινόπωρο στο καλοκαίρι δεν σημαίνει ότι εγώ θα αλλάξω γνώμη. Δεν θα αλλάξω μόδα. Δεν είναι ότι δεν είμαι σε θέση να αλλάξω απόψεις. Αλλά τούτου λεχθέντος έχουμε πολύ σοβαρά προβλήματα τα οποία πρέπει να συζητήσουμε. Έχουμε αυτή τη στιγμή τη συνεδρίαση των G20. Έχουμε αυτά τα οποία ενέκρινε το Συμβούλιο. Έχουμε τις τελευταίες προτάσεις της Κομισιόν από τον Επίτροπο Μπαρνιέ στο Συμβούλιο Κοφίν. Και φυσικά <clears throat> έχουμε και τη μόδα που προέρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες που ζητάν ορισμένα α, χρηματοπιστωτικά εδρήματα που έχουν συστημικό χαρακτήρα να υπόκεινται σε διαφορετική μορφή εποπτείας. Αλλά για να μιλήσουμε για συστημικό φορέα δεν μπορούμε να βαστούμε μοναχά στο μέγεθος. Εγώ συμφωνώ ότι για να προκαλέσει συστημικό χαρακτήρα μια επιχείρηση αυτό έχει να κάνει περισσότερο με τον τρόπο επιχείρηση, με το επιχειρηματικό της μοντέλο, με τη σύνδεση με υποκαταστήματα και θηγατρικές ε, επιχειρήσεις. Είναι διαφορετικό το να έχουμε, να έχουμε στεγανά ε, υποκαταστήματα και θηγατρικές επιχειρήσεις. Δεν είναι το ίδιο να έχουμε μια επενδυτική τράπεζα από ότι να έχουμε μια τράπεζα κλασικού χαρακτήρα. Είναι διαφορετικό να εμπλέκεται κανείς στην αγορά παραγόγων και να έχει χαρτοφυλάκιο συναλλαγών και να μην έχει. Πώς θα επιλύσουμε λοιπόν αυτό το πρόβλημα της πολυπικιλίας. Η Σιλβί Γκουλάρ υποστήριξε δύο επιχείρηματα, τα οποία φαίνεται ότι είναι αντιφατικά μεταξύ τους. Είπε καταρχήν ότι το να θέσουμε ένα φορέα στον κατάλογο των συστημικών φορέων σημαίνει ότι κατά κάποιο τρόπο τον δακτυλοδεικτούμε, αλλά συγχρόνως δίνει και ένα ε, ανταγωνιστικό πλεονέκτημα γιατί θεωρούμε ότι είναι ένας φορέας ο οποίος θα διασωθεί. Αλλά δεν μπορούμε να ακολουθούμε και τις δύο αυτές αντίμαχες απόψεις, κύριε Γουλάρ. Τούτου λεχθέντος. Το πρόβλημα είναι ένα πρόβλημα ουσίας. Όταν υποβάλλουμε ένα φορέα συστημικό, ένα φορέα που δεν μπορούμε να τον αφήσουμε να πτωχεύσει χωρίς να δημιουργήσει προβλήματα για το σύστημα και την οικονομία την πραγματική. Όταν λοιπόν υποβάλλουμε ένα τέτοιο φορέα και λέμε ότι πρέπει να υπόκειται σε ιδιαίτερη υποπτία και όταν ζητάμε από αυτούς τους φορείς να συμβάλλουν σε ένα ταμείο για να μην πληρώνουν την ύφη οι φορολογούμενοι. Αυτό το κάνουμε εκ των υστέρων ή θα πρέπει να δούμε στη συνέχεια αν καλύπτουν ένα σύνολο χαρακτηριστικών που καθορίζουν το ότι είναι συστημικά σημαντικός φορέας. Αν λοιπόν ξεκινήσουμε να λέμε ότι εσύ και εσύ και εσύ είσαστε συστημικοί φορείς, τότε θα έχουμε κάποια προβλήματα. Θα πρέπει λοιπόν να κανονίσουμε αν Αποφασίσουμε εκ των προτέρων ποιοι είναι αυτοί οι φορεί ή αν θα το δούμε επί τη βάση των κριτάρων. Και ένα τελευταίο πρόβλημα το οποίο έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Η ανοιξιατική μόδα έχει περάσει και στα εθνικά κράτη. Γιατί κάποια κράτη-μέλη είπαν ότι θα δημιουργήσουν ταμεία διάσωση. Αλλά α πούμε ότι έχουμε μια γερμανική εταιρεία η οποία έχει ένα υποκατάστημα στην στο Ηνωμένο Βασίλειο, επομένω κάποιο ο οποίο συνεργάζεται με ένα υποκατάστημα γερμανική εταιρεία θα καλύπτεται, αλλά και το ίδιο για κάποιο που λειτουργεί με ένα υποκατάστημα γαλλική εταιρεία. Λοιπόν, θα καλύπτονται σε αυτή την περίπτωση. Αλλά εκεί πέρα πρέπει να δούμε ότι υπάρχει μια στρέβλωση ανταγωνισμού. Εγώ σας υπενθυμίζω το Σαμψόν και τους Φιλιστέους. Όταν ο Σαμψόν βρέθηκε σε μεγάλο κίνδυνο, είπε αποθανέτω η ψυχή μου μετά των άλλων φίλων. Εμείς δεν θέλουμε να βρεθούμε στην κατάσταση των φιλιστέων. Δεν είναι θετικό το να πέσει ένα, <clears throat> ένας ναός στο κεφάλι μας και να πρέπει στη συνέχεια πάλι να δίνουμε λεφτά για να τον ξαναοικοδομήσουμε. Όπως είπε κυρία Φόρτ, υπήρχαν υπάρχει το θέμα του αν θέλουμε να έχουμε ένα ταμείο ή δύο ταμεία. Γιατί δύο ταμεία. Γιατί ο προορισμός είναι διαφορετικός. Άλλο είναι να πληρώσουμε τις παρεμβάσεις για να μην τις πληρώνουν οι φορολογούμενοι και το άλλο ταμείο για την προστασία των καταθετών. Πρέπει λοιπόν να διαχειριστούμε και το επίπεδο των ε, καταθέσεων και το επίπεδο κινδύνου. Γι' αυτό Και η μεγάλη δυσκολία είναι ο λεγόμενος ηθικό κίνδυνος. Γιατί αν ένας φορέας είναι έτοιμος να πτωχεύσει και δεν μπορούμε να τον αφήσουμε να πτωχεύσει γιατί μετά θα πρέπει να πληρώσουν όλοι οι Φιλιστέοι για την διάσωση του ναού και την ανοικοδόμησή του και πρέπει αυτό να γίνει με βάρος των φορολογουμένων, τότε τελικά δίνουμε κάποια μαξιλαράκια σε ορισμένες επιχειρήσεις που δεν τις έχουν όλοι. Από τη μία πλευρά θα υπάρχει λοιπόν η διάσωση, θα υπάρχει η δυνατότητα εκπομπής, <clears throat> να υπάρχει δυνατότητα εκπομπής ε, ε, δανείων που θα τα πληρώνει όλο το σύστημα και σε τελική ανάλυση υπάρχει προσφυγή στους φορολογούμενους. Εμείς δεν θέλουμε να έχουμε μια κατάσταση στην οποία η πραγματική οικονομία πρέπει να πληρώσει για την αποτυχία του χρηματοπιστωτικού συστήματος και επομένως απαιτείται μια προχρηματοδότηση από τον ίδιο τον χρηματοοικονομικό τομέα. Νομίζω ότι εδώ υπάρχει μια συμφωνία, αφάνηκε και στη συμφωνία στη συζήτηση των G20. Οι μόνες χώρες που δεν συμφώνησαν τότε ήταν η Νέα Ισλανδία και ο Καναδάς. Η Νέα Ισλανδία έχει ένα σύστημα που λειτουργεί μέσα από θηγατρικές εταιρείε, οι οποίες υπόκεινται στην εθνική ε, εποπτεία σε ό,τι αφορά τον ανταγωνισμό και τη ρευστότητα και ακολουθεί είναι ένα υπόδειγμα το οποίο είναι αντίθετο από αυτό το οποίο χρησιμοποιείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς έχουμε διαφορετικά συστημικά ιδρύματα, έχουμε διαφορετικά ιδρύματα ευρωπαϊκού χαρακτήρα. Μπορεί να υπάρξει πολύ εύκολα η διάδοση μιας κρίσης σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν και επίπτωση στην πραγματική οικονομία. Επομένω, αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει. Μια τελική παρα μια τελική προειδοποίηση. Αν δεν κάνουμε εμεί κάποια πράγματα τώρα, δεν θα γίνουν ποτέ. Όταν περάσουν τα αποτελέσματα τη κρίση, θα επανέλθουμε στο μοντέλο business as usual, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Εκτό αν έχουμε μια κρίση η οποία θα δημιουργήσει πάλι τεράστιες κρίσεις στην αγορά και τότε μονάχα όταν υπάρξει μια νέα κρίση τότε θα καταλάβουμε αν έχουμε πράγματι φέρει σε, πέρα στις ευθύνες μας. Η μάχη της Αγγλίας κερδίθηκε όταν αποφασίστηκε να αγωνιστεί η Αγγλία κατά της Γερμανίας και όχι όταν τελείωσε η μάχη. Δεν θέλω εγώ να κάνω τον ε, Ισπανό πατριώτη, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ πιο εύκολο να καταλήξουμε σε μια συμφωνία για αυτό το πακέτο με την Ισπανική Προεδρία από ότι με τη Βελγική Προεδρία, τη στιγμή που αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε ποιο θα εκπροσωπεί την Βελγική Προεδρία στα θέματα αυτά. Εγώ πιστεύω λοιπόν ότι είναι απαραίτητο να υπάρξει μια μεγάλη μια ταχύτητα στο βαθμό του δυνατού και θα σας το πω ε, ειλικρινά δεν το λέω αυτό γιατί θέλω να δώσουμε το, την, τον κότεινο του θριάμβου στον κύριο Σαπατέρα αλλά γιατί είναι ο τρόπος με τον οποίο θα μπορέσουμε να διεκπαιρεώσουμε το θέμα αυτό με τον καλύτερο τρόπο. Τώρα αν χρειαστεί να καθυστερήσουμε την ε, ψηφοφορία, εγώ το δέχομαι ότι υπάρχουν θέματα τα οποία είναι πάρα πολύ πολύπλοκα και πρέπει να υπάρξει και η συμφωνία των εισηγητών και φυσικά και των πολιτικών ομάδων στη συνέχεια. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί ένα κοινοβούλιο δημοκρατικό και ανοιχτό. Και εγώ θέλω να συνεχίσω τη συζήτηση αυτή με όλους τους εισηγητές είτε είναι σκιώδες είτε δεν είναι σκιώδες. Uh, thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Δεν το πιστεύω. Τελειώσαμε και δέκα λεπτά νωρίτερα. Α, σανσός. Θα πάει στο λόγο. Δύο λεπτά μονάχα εγώ. Δύο λεπτά μονάχα. Εγώ υποστήριζω αυτά που είπε ο Γκαρσία Μαργκάγιο. Δεν πρόκειται να μπω τώρα στη συζήτηση για τη συστημική εποπτεία. Αυτό είναι ένα από τα σημαντικά προβλήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, αλλά σας λέω και πάλι ότι αυτό δεν αρκεί για να τεκμηριώσει μια καθυστέρηση, γιατί σε μια εβδομάδα θα καταλήξουμε πάλι να είμαστε στην ίδια κατάσταση. Επομένως, είναι το καλύτερο είναι να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη διαδικασία, η οποία θα είναι μακροσκελής βέβαια, και να προχωρήσουμε μέχρι να καταλήξουμε σε μια ψηφοφορία στην Γι' αυτό σας ζητώ να είμαστε όσο δυνατόν ταχύτεροι και καλύτεροι, να ξέρουμε ότι θα πρέπει να είμαστε σε θέση να τηρήσουμε τις ε, υποχρεώσεις μας θα πρέπει μέχρι τον Ιανουάριο να έχουμε κάποια λύση και για τις, για τις εταιρείες πιστοληπτικής αξιολόγησης και να μπορέσουμε να πάμε στην επόμενη συνάντηση των G20 με κάποια λύση ήδη σε ευρωπαϊκό <clears throat> επίπεδο. Εάν δεν υπάρξει κάποιο πρόσκομα λοιπόν θα πρέπει να διατηρήσουμε τις ημερομηνίε που έχουμε καθορίσει τώρα. Αυτό δεν σημαίνει θα λύσουμε όλα τα προβλήματα. Σημαίνει απλώς ότι καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου συζήτησης εμείς θα βελτιώνουμε τις λύσεις μας η Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων είναι τμήμα μια κοινοβουλευτική διαδικασία, αλλά δεν είναι το σύνολο τη κοινοβουλευτική διαδικασία επομένω θα πρέπει να έχουμε μια σωστή διαχείριση του χρόνου. Ευχαριστώ. Τελειώσαμε. Αν κάποιο θέλει να μου μιλήσει, θα μείνω εδώ μερικά λεπτά ακόμα και μετά έχουμε και άλλη συνάντηση το απόγευμα. Τι έχουμε? Έχουμε συνεδρίαση συντονιστών σήμερα.